Συνάδελφοι, αγαπητοί συντονιστές μάλλον, έχετε την αίσθηση ότι έχουν έρθει όλοι οι απαραίτητοι παρόντες στην αίθουσα για να αρχίσουμε την ψηφοφορία, κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να ρωτήσω εσάς και τους συναδέλφους αν όλοι έχετε λάβει τις προφορικές τροπολογίες, τις πιο πρόσφατες. Είναι στο κείμενο, έτσι. Ωραία λοιπόν. Δεν χρειάζεται να τις εξηγήσω τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται να τις αναγνώσετε. Είναι γνωστές. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Τι άποψη έχουν οι συντονιστές. Είναι εδώ όλοι όσοι θα πρέπει να είναι. Αισθάνεστε ασφαλείς. Καλημέρα λοιπόν συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Απλώς προηγουμένως, αν γίνεται, δοκιμάστε τις ε, κάρτες σας να δείτε αν λειτουργούν. Α κάνουμε μια δοκιμή λοιπόν και αρχίζουμε τι ψηφοφορίε. the... Ε, δεν ψήφισαν όλοι. Υπάρχει μια διαφορά ψηφοφόρων και καρτών. Γιωακίμ δεν έχει κάρτα. Οπότε θα πρέπει να προσθέτουμε κάθε φορά τον συνάδελφο. Has... Υποθέτοντας ότι όλοι έχουν ε, την κάρτα τους, εκτός από τον ε, συνάδελφο, θα ξεκινήσουμε με το σημείο 8. Έκθεση της κυρίας Ραμόνα Νικόλ Μανέσκου, χρηστή διακυβέρνηση σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω την αντίποση ότι θέλει να πει κάποια εισαγωγικά σχόλια, κυρία Μανέσκο. Όχι, είναι αυτά που ήδη είπατε. Ωραία. Ενημερωτικά σας λέω ότι έχουμε εδώ 61 τροπολογίες και έχουμε και 7 συμβιβαστικέ τροπολογίες ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεών μας. Λοιπόν, την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 17. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι.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 Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Και υπάρχει και προφορική τροπολογία εδώ. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Ψηφίζουμε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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπάρχει και προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι. Ψηφισμό όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 αποσύρεται. 46 ε, καταπίπτει. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 με προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Ωραία. Ψηφισμό όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι κατάλαβα. 7. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Επτά λοιπόν, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα. Πέρας. 23 υπέρ. Γιάννη, ήσουν υπέρ από ό,τι κατάλαβα. 24 λοιπόν και 9 κατά. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τροπολογία 9 με την προφορική της τροπολογία είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ και ο Γιώχαν. Άρα 35. Όλοι λοιπόν υπέρ είμαστε ομόφωνοι. So I didn't have to say... Δεν χρειάζεται να πω συγχαρητήρια, ήταν πάρα πολύ σαφές. Ο Μιγγέλ λέει ότι από ό,τι θυμάται είναι η πρώτη φορά που έχουμε ομόφωνη ψήφο. Αυτό σημαίνει χρηστή διακυβέρνηση. Μάλιστα. Περνάμε σε κάτι που μπορεί να μην είναι τόσο ομόφωνο. Το ψήφισμα που θα συνοδεύσει την, προσωπική, προφορική μας ερώτηση για την ε, πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική μετά το 2013. Έχουμε τις τροπολογίες 27 ε, και 28. Θα τις ψηφίσουμε ξεχωριστά γιατί δεν υπάρχει συμβιβαστική τροπολογία. Οπότε, ψηφίζουμε. Περνάμε στην τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 αποσύρεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε στη 18 Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε τη 18 πώς τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Okay, they are identical. So, colleagues... Α, είναι ταυτόσιμες οι 19 και 20, οπότε τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται και οι δύο. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Ε, συγγνώμη. Αποσύρθηκε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και για τις αιτιολογικές αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχη ψηφοφορία. De... Πέρας της ψηφοφορίας. Ένας ακόμη και ο Ιωακήμ. Οπότε 39 υπέρ και 31 αποχές. Μάλιστα. Τέλο πάντων, δεν είναι πολύ άσχημα. Περνάμε τώρα στο σημείο 10. Έχουμε εδώ τον κύριο Ιαν Όλσον που είναι ο εισηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ah, Α, έρχεται στις 10. Άμαν, έχουμε πάρα πολύ καιρό, 40 λεπτά. Μήπως μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα σημεία τη ημερήσία διάταξη. Στις 10 έχει προσκληθεί ο κύριος Όλσον, οπότε μπορούμε να περάσουμε στις, στις αποφάσεις που έλαβαν εκθέσεις συντονιστές. Είχαμε το σημείο 1 για την ε, κατανομή των ε, εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων για τις μη νομοθετικές ε, εκθέσεις, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά, την πήραν η ΕΛΚ. Το επόμενο θέμα αφορούσε ε, τις δημοσιονομικές προοπτικές και τις προκλήσεις πολιτικής ε, για την ΑΙΦΟΡ Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Και αυτή την έκθεση την πήραν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ποιος. Και μετά ε, α, αξιοποίηση δυναμικού για τις ε, ε, καινοτόμες επιχειρήσεις. η συντηρητική και η νέα περιφερειακή πολιτική και τουριστική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και πάλι οι σοσιαλιστές. Επίσης υπήρξαν προτάσεις για δημόσιες ακροάσεις. Μικρόφωνο παρακαλώ. Και αποφασίσαμε ότι οι προτεραιότητε για μεγάλες ακροάσεις ε, θα δοθεί στην, ε, στην, ε, έκθεση, στην πολιτική συνοχή, θα χρησιμοποιηθεί η πέμπτη έκθεση συνοχής ως βάση, όπως επίσης και μία ακρόαση για ένα σύστημα προσανατολισμένο περισσότερο προς τους στόχους και τα αποτελέσματα της περιφερειακής πολιτικής και για την πολιτική συλλογή, συνοχής και το ΑΕΠ Για όλα αυτά θα γίνουν ε, σημαντικές ε, μεγάλες ε, δημόσιες ακροάσεις. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που προτάθηκαν θα έχουμε μίνι ακροάσεις. Αλλά δεν θα αποφασίσουμε τώρα τις ημερομηνίε. Επίσης, Περιμένουμε λεπτομέρειες από τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με τις ε, προτάσεις που παρουσιάστηκαν για τις δημόσιες ακροάσεις. Οπότε, ε, σε σχέση με τις αντιπροσωπείες για το 2011 είχαμε επίσης μια ανταλλαγή απόψεων και υπήρξε συμφωνία για το 2011 να προτείνουμε τρεις αντιπροσωπείες, μία στην Ελλάδα, μία στη Γουιάννα και ενδεχομένως και σε άλλες ε, απομακρυσμένες γαλλικές περιοχές. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πολιτικές ομάδες να μας στείλουν ε, ένα ε, προσχέδιο προγράμματος για τις αντιπροσωπείες αυτές, γιατί πρέπει να τις στείλουμε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Οπότε, Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 11, γιατί η κυρία ε, Χιουσμένοβα ήρθε. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Χιουσμένοβα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, το οποίο θα συντάξει για την εφαρμογή της οδηγίας 2623 ε, περί υπηρεσιών θα σας δώσω το λόγο, δεν ε, θα λάβουμε αποφάσεις σήμερα. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κυρία Χιουσμένοβα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το ε, σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την εφαρμογή οδηγίας περιπηρεσιών ε, στην εσωτερική αγορά. Εγκρίθηκε στο τέλος του 2006 και σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν εναρμονίσει την εθνική τους νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Το έγγραφο είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει από την οικονομική και χρηματοπιστωτική ε, κρίση και θα είναι πολύ σημαντική και για τα επόμενα χρόνια για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, ε, την οικονομική ανάπτυξη τη σταθερή, όπως επίσης και τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η οδηγία περί είναι μια εγγύηση για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία ε, μετακίνησης. Επίσης ενθαρρύνει την ισορροπημένη ε, ανάπτυξη, ε, στα, τη σταθερή ανάπτυξη και την συντονισμένη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για κάτι που ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη και τονίζει την σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης για τη σχέση μεταξύ εσωτερικής αγοράς και πολιτικής συνοχής. Το σχέδιο αυτό μας κατευθύνει προς ένα σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και την ενιαία θηρίδα υπό το φως ε, της ε, ε, διαλειτουργικότητας ε, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρώντας τις εγγυήσει για τον περιορισμό των ε, διοικητικών περιορισμών των επιπροσθέτων για τα κράτη-μέλη στηρίζεται η άποψη ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει θετικό ε, αποτέλεσμα και θα υποστηρίξει την ε, οικονομική, ε, δαφική και κοινωνική συνοχή. Υπ' αυτήν την έννοια υπενθυμίζει τη δυνατότητα το, του να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για τη βελτίωση των υποδομών και ε, της ε, πραγματικής ενίσχυσης των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ώστε να αμβληνθούν οι διαφορές μεταξύ τους. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Περχέγγεν για την συνεργασία της στην σύνταξη του παρόντος κειμένου. Ήταν δική της ιδέα να συμπεριλάβουμε την αρχή της πολυγλωσσίας στην ενιαία θηρίδα και ε, την ενίσχυση, την ενθάρρυνση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν μία από τις επίσημες ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεταξύ των αρχών και των παρόχων υπηρεσιών. Επίσης, επιμένουμε στην παρακολούθηση του αντικτύπου της οδηγίας που πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας συγκεκριμένος έλεγχος των περιορισμών σε σχέση με τις υπηρεσίες κοινού οικονομικού ε, ενδιαφέροντος. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που έχω συμπεριλάβει στο κείμενό μου μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψει των συναδέλφων και τις προτάσεις του για την ανάπτυξη του κειμένου με σκοπό να είναι επωφελέ το κείμενο για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Περιμένω τις προτάσεις και τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Χιουσμένοβα. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να πάρετε το λόγο να μας κάνετε, να, μας το επισημάνετε. Με συγχωρείτε. Εγώ Είναι το όνομά μου. Ζήτησα το λόγο διότι είμαι σκιώδης εισηγήτρια των Πρασίνων για το θέμα αυτό και εξετάζουμε το όλο ζήτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ε, στην Επιτροπή αυτή την περασμένη εβδομάδα ήδη εξετάσαμε μια έκθεση που μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι γραφειοκρατικές δυσκολίες της οδηγίας αυτής ιδίω στην Γερμανία επηρεάζονται ζητήματα όπως η διοργάνωση των καράζ αυτοκινήτων μέχρι και των ε, νεκροταφείων. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την υλοποίηση της οδηγίας αυτής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις συνέπειες ε, επιλεκτικά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια προσεκτική εξέταση βάσει της εθνικής νομοθεσίας και να φροντίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω διοικητικό άχθος. Ο σκοπό μα είναι να διευκολύνουμε τα πράγματα, όχι να τα δυσκολέψουμε. Πρόεδρο, ε, συνάδελφοι, παρακαλούμε να είστε σαφεί όταν ζητάτε το λόγο. Κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, την για την πρόταση αυτή και θα συμφωνήσω με τα σχόλια της κυρίας Ρούλε όταν λέει ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε υπερβολικό διοικητικό άχθο και ότι θα έχουμε πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την πρόταση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί και τι όχι. Θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα στο σημείο 4 σε ό,τι αφορά τις διοικητικές ε, υπηρεσίες, φαίνεται εδώ να υπάρχει η άποψη ότι κάποιες ε, δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να εισάγουν πολυγλωσσικές ε, υπηρεσίες. Αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Βεβαίως από τις πιο ισχυρές δημοτικές αρχές καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ενσωματωθούν όλοι οι πολίτε με διαφορετικέ γλωσσικέ ανάγκε. Αλλά να τα πετύσουμε αυτό από όλε τι δημοτικέ αρχέ μου φαίνεται ανέφικτο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να εκφράσουμε αυτή την ιδέα διαφορετικά, ίσω δίνοντα κάποια ενθάρρυνση, παροτρύνοντα τι δημοτικέ αρχέ υπό το φω τη παγκοσμιοποίηση, να προσπαθήσουν να διευκολύνουν τα καθήκοντα όσων χρησιμοποιούν διαφορετικέ γλώσσε. Αλλά δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε. Από ό,τι βλέπω, δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο. Όχι. Παρακαλώ. Zunächst einmal entschuldigen, dass ich zu spät war. Wir hatten noch Abstimmungen auch im Kulturausschuss als äh, Schattenberichterstatterin für die EVP. Με συγχωρείτε για την ε, καθυστερημένη αφήξή μου. Βρισκόμουν σε άλλη επιτροπή. Ω και για το ΕΛΚ, να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το σχέδιο αυτό έκθεση. Όμω, όπω και η κυρία Κρέιλ, θα ήθελα και εγώ να σταθώ σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Ήδη το έχω αναφέρει και έχω καταστήσει σαφέ ότι η πολυγλωσία στι ενιαίε θηρίδε είναι κάτι μάλλον ανέφετο. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα σε κάθε περίπτωση. Μάλλον τα αγγλικά. Στις ενιαίε θηρίδε όμως να ισχύει αυτό και μόνο και όχι στις δημοτικές αρχές διασυνοριακά, διότι αλλιώ θα προκαλέσουμε τεράστιο διοικητικό άχθο για τις τοπικές αρχές και αυτό θα δυσκολεύσει τις τοπικές κυβερνήσεις των κρατών μελών. Θα ήταν πραγματικά υπερβολική απέτηση αυτή. Κατά συνέπεια, προτείνω αντί να παραμένουμε στι τρει επίσημε γλώσσε, όπω αναφέρεται, να ζητήσουμε την πρόθεση των επισήμων γλωσσών που τουλάχιστον ομιλούνται στα γειτονικά κράτη. Δηλαδή, τα αγγλικά να είναι η lingua franca, η γλώσσα συνεννόησης, η διεθνής, και μια επιπλέον για κάποιες άλλες περιοχές. Στη δική μου περίπτωση, λόγω χάρη, θα μπορούσαν να είναι τα γαλλικά ή τα ολλανδικά, στην περιοχή από την οποία προέρχομαι. Για να διευκολύνουμε τις δυσυνοριακές επαφές σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Νομίζω ότι έτσι θα διευκολύνουμε αρκετά τη ζωή μας ε, κατά την διοργάνωση των ενιαίων θηρίδων. Μια επιλογή λοιπόν θα ήταν να προκρίνουμε τα αγγλικά και βεβαίως να είναι υποχρεωτική και η μετρική γλώσσα της κάθε χώρας. Κατά τη δική μου άποψη τα αγγλικά είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη επιλογή. Και μια άλλη επισήμανση. Η υποχρεωτική κοινοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στα καταστατικά μέχρι τώρα αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι οποιαδήποτε αλλαγή να κοινοποιείται στις τοπικές αρχές. Και αυτό προκαλεί τεράστιο διοικητικό άχθος. Στα πλαίσια όμως της υλοποίησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η υλοποίηση της συστηματικής κοινοποίησης. εάν κάθε αλλαγή στο καταστατικό πρέπει να ε, κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε κλιμάκιο των δημοτικών αρχών, αυτό εκπροσωπεί ένα τεράστιο φόρτο εργασία. Ιδίω σε μια παρόμοια διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να κοινοποιηθούν οι ανάλογε αλλαγέ και στην Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι επικοδομητικό να επιμείνει σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ιωάχιμ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μας έχουν λίγο ξεπεράσει τα γεγονότα. Η οδηγία υπηρεσιών έπρεπε να έχει αρχίσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2010. Εμένα θα με ενδιαφέρε περισσότερο να ακούσω λίγο περισσότερο τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη τι ακριβώς ε, ζητούμε εδώ, γιατί επηρεάζεται μία διαδικασία που έχει ήδη δρομολογηθεί και ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν αλλαγές. Θέλουμε να εναρμονίσουμε περαιτέρω ό,τι έχει γίνει ως τώρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε τις ε, τοπικές αρχές τι χρειάζονται, τι ακριβώς επιθυμούμε όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της εφαρμογής ε, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, είναι ζήτημα κράτους μέλους και δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι γίνεται πλήρης εφαρμογή των διατάξεων ε, στα, σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις αυτές. Θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε το άχθος ε, στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές που ε, ήδη έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Νομίζω <coughs> ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποτε η θεωρία να συναντήσει την πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούλα θέλει να πάρει το λόγο. Ναι. Μπορώ να είμαι σύντομη. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, είναι αρμόδια για την ε, έκθεση αυτή. Συνήθως μετά την εφαρμογή αρχίζουμε, ε, περνούμε σε μια αξιολόγηση. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι η συγγήτρια και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε προβλήματα στην εφαρμογή. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, έχουν να κάνουν ε, με τις συνθήκες ε, στα κράτη-μέλη που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της οδηγίας ή έχει να κάνει με την παρακολούθηση της εφαρμογής που είναι επίσης κάτι το πολύ σημαντικό. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία και αυτό δεν το θέλει κανείς, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, Νομίζω ότι οι προτάσεις μου έχουν να κάνουν με ολόκληρη την εφαρμογή του κειμένου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Χιουσμένεβα, θέλετε να απαντήσετε. Аз Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους. Εγώ είχα ήδη μια ανταλλαγή απόψεων με κάποιους από εσά ε, πριν από τη συνεδρίαση, κατά τις τελευταίες εβδομάδες και νομίζω ότι εντός της ε, προθεσμίας ε, για τις τροπολογίες οι σκιώδεις εισηγητές τουλάχιστον θα είναι σε θέση να υποβάλουν ε, επισήμως τις προτάσεις τους, ώστε το τελικό σχέδιο γνωμοδότησης ε, να μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Ενδεχομένως ε, η συνάδελφος να άργησε, αλλά εγώ είπα στην εισαγωγή μου ότι κάποιες από τις τροπολογίες τις έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο πρώτο σχέδιο του εγγράφου μου και βέβαια θα ήθελα να καθησυχάσω τους συναδέλφους ότι οι προτάσεις τους και κυρίως αυτές της γερμανικής αντιπροσωπείας θα συμπεριληφθούν επίσης. Μάλιστα. Έχει γίνει αναβολή της έκθεσης από την ε, Επιτροπή της ε, Εσωτερικής Αγοράς κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τον ε, Ιανουάριο. Τον Οκτώβριο θα ξέρουμε κατά πόσο θα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη τον Οκτώβριο για να ανοίξουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα ήθελα να καλέσω τους κοιόδης εισηγητές να συνεργαστούν με την κυρία Χιουσμένοβα ώστε να καταλήξουμε σε μία ε, αποδεκτή γνωμοδότηση. Ο κύριος Όλσον είναι πλέον μαζί μας. Μπορούμε να πάμε πίσω στο σημείο 10 ο κύριος Γιάνν Όλσον είναι ο εισηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε σχέση με έκθεση που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματική εταιρική σχέση στην πολιτική για τη συνοχή. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να σας πω το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Ήταν αίτημα του κυρίου Σπίτλα και της κυρίας Χουβνέρ ε, στην προηγούμενη ε, σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν λοιπόν και εσείς υπεύθυνοι. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, λέει η κυρία Χουβνέρ Όχι, λέει ο κύριος Όλσον, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ σωστό το αίτημά σας και αφορούσε την εξέταση της ε, ε, αρχής ε, της εταιρικής σχέσης, ειδικότερα όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, η οικονομική κοινωνική εταίροι, οι κυβερνητικές οργανώσεις, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η κοινωνική οικονομία, ως σκοπό είχαν τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών της αρχής αυτής της εταιρικής σχέσης γιατί αυτό θα αποτελούσε τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελλοντική ε, συνοχή, για τη μελλοντική πολιτική συνοχής σε σχέση με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ε, εταιρική αυτή σχέση. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν τα κράτη-μέλη τη σημασία των εταιρικών αυτών σχέσεων, των συμπράξεων Είχαμε απόψεις από τους κλάδους, από τις περιφέρειες, από τους οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάναμε πολλές επιτόπου επισκέψει ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Και πρέπει να πω ότι είναι μια γνωμοδότηση η οποία πραγματικά ήταν αποτέλεσμα εταιρική σχέση ε, συνεργασίας με τους διάφορους ε, εμπλεκομένους φορείς. Βέβαια είναι κάτι το οποίο έχετε συζητήσει πολλές φορές και γνωρίζετε γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Απλώς θα ήθελα εντάχει να πω ότι αφορά μία πραγματική εις βάθος συνεργασία η οποία μπορεί να βελτιώσει ε, την ε, συνοχή. Χρειάζεται ισότιμη συμμετοχή των ιδιωτικών ε, εταίρων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σωστά και να είναι ενεργός η συμμετοχή τους. Η αρχή αυτή τη εταιρική σχέσης σημαίνει επίσης ότι οι τοπικοί φορείς, οι ανάγκες των τοπικών φορέων ε, θα εξυπηρετηθούν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και ενισχύεται έτσι η συνεργασία μαζί τους, ε, υπάρχει μεγαλύτερη σχέση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων φορέων, δηλαδή μέσω της αρχής αυτής ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται πραγματικά σε τοπικό επίπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Η... Το να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ιδιωτικοί εμπλεκόμενοι φορείς είναι μια κατάσταση επικερδής για όλους. Τα γενικά συμπεράσματα στην έκθεση είναι ότι το άρθρο 11 πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 11 του Γενικού Κανονισμού που ξέρετε ότι είναι αυτό που ορίζει την αρχή της εταιρικής ε, ε, σχέσης. Δεν θέλουμε όμως ε, να δοθεί πολύ μεγάλο περιθώριο για εθνική ερμηνεία της αρχής της εταιρικής σχέσης και εμείς προτείναμε στην έκθεσή μας αλλαγές διατύπωσης στο άρθρο 11. Ένα δεύτερο, Ένα δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι πιο ενεργός, πιο δραστήριος σε σχέση με την αρχή αυτή. Γιατί είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο παρακολουθούσε, ε, ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία, αλλά δεν συμμετείχε τόσο ενεργά στην πολιτική συνοχή όπω το παρελθόν. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι οι εθνικέ νοοτροπίε πρέπει να αλλάξουν, ακόμη και για την ε, διάδοση των ε, καλύτερων πρακτικών. Η διάδοση αυτή μπορεί να, ήταν, να είναι πολύ αποτελεσματική, πιστεύουμε, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς πρέπει να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον για να είναι αποτελεσματική η αρχή της ε, σύμπραξής τους. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν ε, πόροι τεχνικής ενίσχυσης για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι άκουσα στις επαφές μου με τους διάφορους φορείς, η ανάπτυξη υποδομών είναι ένας πραγματικός ε, όρος για μια αποτελεσματική σύμπραξη. Και τέλος, υπάρχει μια σαφή σχέση μεταξύ της διάρθρωσης του προγράμματος και της ε, σύμπραξης. Όταν η δομή του προγράμματος είναι περισσότερο εστιασμένη, καλύτερα εστιασμένη, υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες σύμπραξης και είναι επίσης ε, πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα της σύμπραξης αυτής. Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να βασιζόμαστε στις καλύτερες πρακτικές. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Έχουμε και παραδείγματα κακών πρακτικών βεβαίως, αλλά οι καλές πρακτικές, οι καλύτερες πρακτικές είναι πολλές. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, η σύμπραξη αυτή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι συστηματική. Έχει ενσωματωθεί στο, στην αγγλική περιφερειακή πολιτική, στη διάρθρωσή της. Και μια πραγματική και μοναδική περίπτωση είναι το πρόγραμμα της Ισπανίας. Γιατί υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι οι ίδιοι οι εταίροι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του προγράμματος. Επίσης, κοινωνική εταίροι για ανάπτυξη υποδομών. Είναι κάτι που συμβαίνει και στην Νότια Ιταλία. Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα και η Νότια Ιταλία. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το πρόγραμμα ποιής όπου οι, ε, οι πολιτικές ε, είναι ολοκληρωμένος, ε, ολοκληρωμένες, δηλαδή αξιοποιούνται όλοι οι πόροι που υπάρχουν και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο με, αποκεντρωμε... με αποκεντρωμένο τρόπο. Υπάρχει δηλαδή διαχείριση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των πόρων. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η Αυστρία. Με ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στα τέλη της ε, δεκαετίας του 80. Οι επιδοτήσεις αποδείχθηκαν ε, πάρα πολύ σημαντικές. Το Ίσπρα, για παράδειγμα, το Σκάνι στην Ιταλία, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και υπάρχει και το παράδειγμα της Γαλλίας, όταν δηλαδή δόθηκαν επιδοτήσεις ειδικότερα σε τοπικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους. Μπορούν δηλαδή από μόνε του οι εταιρείε μετά να διαχειρίζονται του πόρου του, ε, να συμμετέχουν σε ευρύτερα προγράμματα κλπ. Και κάτι ακόμη. Στην Πολωνία υπάρχει αυτό το πρόγραμμα αποκεντρωμένη διαχείριση. Ε, είναι υπεύθυνη διαχείριση τη δική του περιφερειακή ε, ανάπτυξη, πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη. Κάτι που τους δίνει πολύ σημαντικό για την Πολωνία. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τις βασικές μας συστάσεις. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσει ε, για την ύπαρξη σύμπραξης. Το άρθρο 11 βέβαια είναι ένα βασικό άρθρο, αλλά θα έπρεπε να αναπτυχθεί επίσης ένας ε, κώδικας ε, καλύτερων πρακτικών. Έχουμε κατευθυντηρίες γραμμές ε, που πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη ή που πρέπει να αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Και είναι κάτι που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε περαιτέρω την ιδέα αυτή της σύμπραξης. Ή τα ολοκληρωμένα και στοχευμένα προγράμματα. Στόχος, πεδίο εφαρμογής. Νομίζω ότι για αυτά τουλάχιστον θα ενισχυθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης ε, και ζητούμε κάποιες κοινοτικές πρωτοβουλίες ε, να επιστρέψουν ε, επιδοτήσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάποια από αυτά τη χρησιμοποιούν ήδη, ε, κάποια όμως όχι. Και μια διαδικασία απλοποίησης ε, των πληρωμών. Νομίζω ότι αυτό είναι κάποιο, ένα σχόλιο που το ακούσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη, από όλους τους εταίρους μας. Είναι μια πολύ μακρόχρονη διαδικασία, είναι πολύ χρονοβόρα, περνάει πολύ, χρόνο πολύς χρόνος πριν από την καταβολή των πληρωμών και ακόμη και αν υπήρξε ήδη απλοποίηση χρειάζεται ακόμη περισσότερη. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με τη διάρθρωση του προγράμματος. Επίσης, οι περιφέρειες που τα καταφέρνουν καλά θα έπρεπε να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο αριστείας για να μπορούν να διαδίδουν τις ε, βέλτιστες πρακτικές με τον καλύτερο τρόπο. Και τέλος βλέπετε κάποιες σκέψεις ε, για μετά το 2014. Βέβαια είναι κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό τώρα. Αυτό που επιθυμούμε Είναι ολοκληρωμένα προγράμματα, ε, εστιασμένα περισσότερο, στοχευμένα καλύτερα, ακόμη και από γεωγραφικής απόψεως, ε, καλύτερη δηλαδή γεωγραφική κατανομή τους, ε, συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή, συγκεκριμένη αποστολή, πρωτοβουλίες της κοινότητας, τοπική ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τοπική ιδιωτικοί εταίροι να μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον επόμενο κύκλο προγραμματισμού. Very efficient uh, they could be uh, if they used. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, νομίζω ότι είπα τα περισσότερα. Θα προτιμούσα να ολοκληρώσω εδώ για να ακούσω και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Να Ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και την όλη συζήτηση. Ο κύριος Λάστρα, ευχαριστώ. Δεν περίμενα να πάρω το λόγο πρώτος, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι το πνεύμα. Συμμερίζομαι κατά πολύ το πνεύμα της έκθεσης αυτής λοιπόν, διότι είναι σημαντικό για την κοινωνία των πολιτών και όχι μόνο για τους παραδοσιακούς φορείς, αλλά για το άνοιγμα του τομέα αυτού στην κοινωνία των πολιτών ευρύτερα, ώστε να έχουμε αυτή τη διακυβέρνηση και καλή διαχείριση των κονδυλίων θα έχουμε κάνει σε αυτή την περίπτωση ένα βήμα προόδου και θα συμφωνήσω με οποιαδήποτε πρόβλεψη για τεχνικά μέτρα, διότι πραγματικά θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή τη διάσταση. Και θα πρέπει να εξοπλίσουμε την κοινωνία των πολιτών με τα μέσα που θα τις επιτρέπουν να εργάζεται αποτελεσματικά και θετικά στο πλαίσιο όλων αυτών των προγραμμάτων, κατά τρόπο αποτελεσματικό διότι αυτά που περιέχει η γνωμοδότηση αυτή αφορούν ακριβώς τη χρηστή διακυβέρνηση, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όταν λοιπόν εδώ βλέπουμε να υπάρχει βαθιά διασύνδεση των διαφόρων τομέων, αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα από κοινού θα αντιμετωπίζονται καλύτερα και χέρι με χέρι θα συνεργαζόμαστε με τους πολίτες ώστε να λύνουμε τα δικά τους τα προβλήματα και μαζί τους να καλύπτουμε τις ε, ανησυχίες και μεριμνές τους. Όπως λέει λοιπόν ε, η έκθεση αυτή, έχουμε το πρόγραμμα Leader, το πρόγραμμα Urban 2 και στα 27 κράτη-μέλη έχουμε διαφορετικούς τρόπους εργασίας, διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές σχέσεις με τις ενώσεις τους ε, εταίρους μας. Θα πρέπει ενδεχομένως λοιπόν να επεξεργαστούμε κοινέ γενικές αρχές ε, για, σχετικά με, με τις καλύτερες πρακτικές. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ομοιογενή προσέγγιση της ε, κοινωνίας των πολιτών. σημεριζουμε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει ενεργότερη δράση. Πράγματι είναι σημαντικό αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι και το τονίζουμε και στη σχετική και στην ε, λογοέκθεση. Επιτρέψτε μου επίσης να σας συγχαρώ για τη σύνταξη της ε, γνωμοδότησής σας και να πω ότι στηρίζω όλες σας τις πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την αριστεία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, θα πρέπει πράγματι όλες οι περιφέρειες και οι επαρχίες να μπορούν να υποφεληθούν από τις καλύτερες πρακτικές. Όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα βήμα πρόοδου στα πλαίσια της μελλοντική μας πολιτικής συνοχής. Θέλουμε αυτή η πολιτική να είναι πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, πιο δραστήρια. Πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά, διότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους δημάρχους, με τις δημοτικές αρχές για να υλοποιήσουμε προγράμματα, θα μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τέτοιου είδους προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ ξανά για την σύνταξη της σας. Ευχαριστούμε κυρία Σρέτερ. Και μετά ο κύριος Όρο, κύριος Κέλλη κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε την δυνατότητα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό επανελειμμένως. Και χάρη στις ανοιχτές ημέρες, αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ καλές αφορμές για να έχουμε ανταλλαγή υπόψεων και ήταν και πολύ επιτυχημένη η συγκεκριμένη τελευταία μας εκδήλωση. Έχω κάποια ερωτήματα τώρα. Είπατε κύριε Όλσον ότι στο άρθρο 11 πρέπει να επιφερθούν βελτιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, πού ακριβώς πρέπει να γίνουν οι βελτιώσεις και τι θα πρέπει να λέμε. Με τι διατύπωση. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Έπειτα δεύτερο ερώτημα. Είπατε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει απλούστευση στο σύστημα πληρωμών, στι διαδικασίε πληρωμών. Θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο για να πετύχουν περισσότερο οι εταιρικέ μα σχέσει. Σε αυτή την περίπτωση όμω θα χρειαστεί έλεγχο και επαλήθευση του αν ε, σωστά καταβλήθηκαν ε, τα λόγω ποσά. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να προσπαθήσει να ενοποιήσει κάποια συστήματα, τα οποία όμω φαίνεται για την ώρα να είναι αρκετά περίπλοκα και ίσω και πολύ επικεντρωμένα σε κάποιε περιπτώσει. Ποια θεωρείτε λοιπόν εσεί ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα ώστε να μπορούμε και εμεί να προετοιμαστούμε για να διευκολύνουμε το έργο τη Επιτροπή. Και τρίτο ερώτημα. Για τα δίκτυα. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα σα για τα δίκτυα και πιστεύω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο σημείο αυτό για να συγκεκριμενοποιήσουμε τι προτάσει σα. Κύριε Ορό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, ήθελα να σχολιάσω το θέμα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Νομίζω ότι αυτά τα άτομα έχουν περισσότερο ανάγκη από όλου από την αλληλεγγύη μας. Όμως, συχνά η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία έχουν σχέση και με ντορές, άρα με στήριξη. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν θα αποτίσω φοροτιμή στην αφοσίωση όσων ασχολούνται με τα άτομα αυτά. Και εδώ μιλάμε για ανάγκες και οικονομικές, ε, αλλά όχι μόνον. Πολλές φορές μιλάμε για ανάγκες τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των ενώσεων των ατόμων αυτών. Η εύρυθμη λειτουργία των ενώσεων ή των συλλόγων, ιδίω όταν ε, αυτοί οι αυτές λαμβάνουν ε, δημόσια χρηματοδότηση. Οι κανόνε που διέπουν τη λειτουργία του σε αυτέ τι περιπτώσει είναι πολύ αυστηροί και πολύ συγκεκριμένοι. Ξεπερνούν κάποιες φορές τις δυνατότητες των ε, υπευθύνων των ενώσεων και των συλλόγων. Ξέρω λοιπόν ότι σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και το ερώτημά μου, κύριε Όλσον, είναι πώ μπορούμε να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό ποιο είναι το πεδίο παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ιδίω σε ό,τι αφορά τι ανάγκε και τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος ε, θα συμφωνούσε με τα βασικά στοιχεία της παρουσίαση του κυρίου Όλσον. Προφανώ η ανάπτυξη του κώδικα πρακτικής, ε, η απλοποίηση των ε, πληρωμών και η διάδοση των καλών πρακτικών είναι ό,τι καλύτερο. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό. σε κάθε συζήτησή μας συζητούμε κάθε φορά το θέμα της απλοποίησης. Ο κύριος Μπαρόζο το ανέφερε επίσης ε, ε, μια φορά σε κάποια επίσκεψή του και η μείωση του, της γραφειοκρατίας κατά 25% είναι αξιέπαινο στόχος. Αλλά πώς θα το κάνουμε και ποιος θα το κάνει κυρίως. Γιατί εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ καλά προγράμματα και μετά όταν ζήγησαν το κόστος και το χρόνο για την εφαρμογή, τελικά δεν άξιζε το κόπο να περάσουν στην εφαρμογή. Τι θα κάνουμε λοιπόν, νομίζω ότι ο προλαλήστας συνάδελφος ε, μίλησε για τον εντοπισμό των εμποδίων. Πού βρίσκονται αυτά τα εμπόδια, είναι όλα σφάλμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή είναι το ζήτημα θέμα και των κρατών μελών που είναι υπερβολικά ενθουσιώδη, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα στην πράξη. Μήπως θα έπρεπε να συντάξουμε έναν κατάλογο των, των, των στόχων που πρέπει να επιτύχουμε, έναν προς ένα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον απότερό μας στόχο. Τότε νομίζω θα δώσουμε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα είμαστε νομίζω πολύ πιο κατάλληλοι, πολύ πιο σχετικοί στη δουλειά μας ε, και πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με, το, με αυτά που κάνουμε σήμερα. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Όλσον, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε. Ναι, θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας προς την γνωμοδότησή μου, καταρχάς. Διακόπτη Πρόεδρος, έχουμε ακόμη έναν ομιλητή που θέλει να πάρει το λόγο. Σας πειράζει να του δώσω το λόγο πριν απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη σε σχέση με την απλοποίηση. Εγώ είμαι 100% υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σήμερα το ποσοστό ε, αξιοποίησης των ε, πιστώσεων, ε, των, της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής είναι πάρα πολύ χαμηλό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Δεν θα ήθελα μια κακή αξιοποίηση των πόρων αυτών ε, να δημιουργήσει πρόβλημα ε, στην συζήτηση που θα κάνουμε για τον προϋπολογισμό. Κάθε αξιοποίηση πόρων είναι χαμηλή γιατί οι διαδικασίες ε, είναι πολύ περίπλοκες νομίζω και έχω την εντύπωση ότι αλλάζουμε τις διαδικασίες σε κάθε οικονομικό προγραμματισμό και νομίζω ότι αυτό προσθέτει στο περίπλοκο. Γιατί αν σε κάθε οικονομικό προγραμματισμό οι κανόνε του παιχνιδού είναι διαφορετικοί, για τα κράτη-μέλη η εφαρμογή του σημαίνει τροποποιήσει, μεγαλύτερη γραφειοκρατία και περιπλέκει ακόμη περισσότερο την έναρξη τη διαδικασία. Όταν ε, αντί λοιπόν να απλοποιήσουμε, ουσιαστικά περιπλέκουμε τα πράγματα. Αυτό που θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να απλοποιούμε με καλύτερο τρόπο να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε σε πιο μακροπρόθεσμους, ε, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Να έχουμε δηλαδή μία πιο ε, μακροπρόθεσμη διαδικασία και νομίζω ότι τότε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα κύριε Όλσον έχετε πράγματι το λόγο. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω αμέσως στις απαντήσεις των ερωτήσεων. Για το άρθρο 11 στην έκθεσή μου έχω συμπεριλάβει τις αλλαγές που προτείνουμε στο άρθρο 11. Θα το δείτε στο τελευταίο τμήμα της έκθεσής μας, ε, κυρία Σρότερ. Αν, αναδιατύπωση ζητούμε. Δηλαδή, όταν λέει όπου χρειάζεται ή όταν συνάδει με, τους ε, εθνικούς ε, νόμου, με την εθνική νομοθεσία και τις, ε, τους, και τους, τις συνήθεις πρακτικές του κράτους μέλους να λέει και με τη συμφωνία των εταίρων. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό ε, κατευθυντήριες γραμμές και στόχους ε, την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών ε, και την ενίσχυση των βασικών ε, στοιχείων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτή είναι μία έκθεση, μία πρόταση, συγγνώμη, που την έχω αντιγράψει από τη συνθήκη αφορά τον, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο είδους ε, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για να μπορέσει να εφαρμοστεί καλύτερα αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι κακή ιδέα. Επίση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε σε συνεργασία με του ε, εμπλεκόμενου φορεί να έχει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθή Πρακτική για την ε, εφαρμογή τη αρχή αυτή. Κάτι πιο συγκεκριμένο, τέλο πάντων, ε, πέρα από την απλή παρακολούθηση. Αυτά για, τα, για τι αλλαγέ στο άρθρο 11. Τώρα, για το δίκτυο περιφερειών αριστεία. Οι περιφέρειες που θεωρούν ότι είναι οι καλύτερες θα έπρεπε να ιδρύσουν ένα δίκτυο και να ενημερώνουν τις υπόλοιπες περιφέρειες για το πώς ε, θα μπορούσε να, αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν καλύτερα οι προσπάθειες αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι βέβαια που πρέπει να συζητήσουμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών την ίδια. Όσον αφορά την απλοποίηση, πολλοί συνάδελφοι, ο κύριος Κέλλη και πολλοί άλλοι μίλησαν για το θέμα αυτό ε, και η κυρία Οκονή μίλησε για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, είναι κάτι, ένα, ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο συνεχώς προκύπτει ότι είναι περίπλοκες, πολύ γραφειοκρατικές οι διαδικασίες, ε, ότι είναι κάτι το οποίο ανατρέπει κατά κάποιο τρόπο, παρακολεί την αξιοποίηση των ε, ε, διαρθρωτικών κονδυλίων και αποθαρρύνει τον κόσμο από τη χρήση των κονδυλίων αυτών, γιατί είναι πολύ χαρτούρα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Ένας τρο, τρόπος, χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες για την απλοποίηση, και σε πολλές ε, διοικητικέ ε, διαδικασίε είναι να χρησιμοποιούνται για παράδειγμα οι συνολικέ επιδοτήσει. Γιατί τότε θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ε, για μικρότερα προγράμματα, για μικρότερους οργανισμούς Και πράγματι η συνολική επιδότηση δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έρθει σε επαφή από μόνος του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι είναι κάτι πιο εύχριστο Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός ε, ολόκληρη τη διαδικασία και τη προχρηματοδότηση και τη καταβολή των πληρωμών. Ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στι ανάγκε των δικαιούχων, ειδικότερα όταν μιλάμε για μικρότερου φορεί. Εκεί υπάρχει πραγματική ανάγκη και πιστεύουμε ότι εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη μεγαλύτερης προχρηματοδότησης όταν μιλάμε για τους μικρότερους ε, φορείς. Αυτά τα μέτρα ε, πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Οι οργανισμοί που εκπροσωπούν ε, μικρές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινωνικών ε, εταίρων. Ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαδραματίζουν σημαντικό λόγο, ε, ρόλο συγγνώμη, στις εταιρικές σχέσεις, γιατί γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση και γνωρίζουν τι αλλαγές πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και το πώς μπορούμε να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό την ιδέα των ε, διαρθρωτικών κονδυλίων. Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο μίλησα για το καλό παράδειγμα της Ισπανίας, ε, γιατί οι ίδιοι οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του προγράμματος ε, και όπως επίσης και άλλα ιδιωτικά ιδρύματα στην Ισπανία. Είναι πραγματικά επικεντρωμένη και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και έτσι υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες ε, και των διαρθρωτικών κονδυλίων. Γιατί υπάρχει ακριβώς ένα πρόγραμμα που συνδέει τους ε, δύο αυτούς πόλους. Και υπάρχει στην Ισπανία κάτι τέτοιο που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αποκέντρωσης ε, των επιχειρησιακών προγραμμάτων. για να είναι πιο γνωστά, να συζητιούνται περισσότερο και να είναι η διάδοσή τους ε, καλύτερη σε τοπικό επίπεδο. Και γιατί όπως είπα, η πολιτική συνοχής είναι το σημείο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συναντήσει τον πολίτη και πρέπει να προσαρμόσουμε τα εργαλεία ε, διάδοσης της ε, αρχής εταιρικής σχέσης ε, με τέτοιο τρόπο στις πολιτικές, ώστε να μπορούν πραγματικά να είναι προσαρμοσμένα στην ανάγκη, στις ανάγκες των πολιτών και πρέπει τα προγράμματα να είναι διαρθρωμένα με τον κατάλληλο τρόπο. Ε, υπάρχουν επίσης πολύ καλά ε, παραδείγματα τεχνικής αρρωγής ε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, να σας υπενθυμίσω την Ουαλία, τη Σλοβενία επίσης. Η Γερμανία έχει τέτοιου είδους πρόγραμμα. Υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ των οργανισμών που λαμβάνουν τεχνική αρρωγή με σκοπό να γίνει καλύτερη διάδοση των διαρθρωτικών κονδυλίων στην περιφέρεια ή και σε ολόκληρη τη χώρα. Και νομίζω ότι μπορούμε να εμπνευστούμε από τα παραδείγματα αυτά. Από όλε αυτέ τι περιπτώσει δηλαδή, όπου υπάρχει τεχνική αρρωγή, υπάρχει ανάπτυξη ικανοτήτων ε, ε, για τον ιδιωτικό τομέα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ κυρία Όλσον. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η έκθεσή σας για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο νομοθετικό πακέτο το οποίο επεξεργαζόμαστε γύρω από αυτό το θέμα και εμείς είμαστε υπέρμαχοι των πρωτοβουλειών από κάτω προς τα πάνω. Και ελπίζουμε ότι κάτι σαν το Leader, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ε, εποφελές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναδειχθεί περισσότερο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ένα, μία από τις βασικές προκλήσεις ε, είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, γιατί θυμάμαι πολλές φορές ε, εταίρους ε, που υπάρχουν, αλλά η, η παρουσία τους δεν είναι επαρκής γιατί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες εταιρικής σχέσης που τους δίδονται. Επομένως, πρέπει να ε, τους καταστήσουμε ικανούς να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Από ό,τι κατάλαβα έχετε επαφές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να μπορέσετε να επηρεάσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Ο Ζων Πολ είναι μαζί μας. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 12, ΑΕΠ και πέρα από αυτό. Μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπεσέ, που είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης και ποιος ε, συνάδελφος ε, θέλει να λάβει το λόγο μετά, ευπρόσδεκτο. Έχετε το λόγο κύριε Μπεσέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σα στην μεγάλη σημασία αυτή της νομοδότηση που υποβάλλουμε εν ώψη της προτάσεως, μάλλον της ανακοινώσεως της Επιτροπής για τους δείκτες ή τα μέτρα υπολογισμού της πρόοδου. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι στατιστικό δηλαδή μόνο το θέμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό, κεντρική σημασία κατά την άποψή μου ζήτημα. Και γιατί, διότι προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καθοδηγήσουμε για το μέλλον τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολιτικές της περιφερειακής συνοχής. Για την γνωμοδότηση που έχω να υποβάλω στην Επιτροπή μας, προς έγκριση, έχω να πω ότι στόχος της είναι να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής και τις δραστηριότητες της Eurostat, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα σύνολο δικτών επί του ΑΕΠ μέσα υπολογισμού συμπληρωματικά ως προς το μέσον το οποίο τώρα κυριαρχεί, δηλαδή το ΑΕΠ. Αυτά τα νέα μέσα Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν θα έχουμε το κόστος με υπολογισμό δύο δικτών εξωτερικών, δηλαδή περιβάλλοντος και κοινωνικής ενσωμάτωσης, του κόστους της κοινωνικής ενσωμάτωσης ή της κοινωνικής ενσωμάτωσης ως κόστους. Και αυτό σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με όλες τις ε, δραστηριότητες ή τους τομείς, σημαίνει ότι θα έχουμε σε θέση μας μέσα που θα μας εξασφαλίσουν μια καλύτερη γνώση της πραγματικότητας, ε, βέλτιστη αξιολόγηση των καταστάσεων και πιο εύστοχες επιλογές. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή πολιτική θα έρθει πιο κοντά στις ανησυχίες, ανάγκες, προσδοκίες των πολιτών και ιδιαίτερα όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική. διαφορετικά τα μέτρα που θα εισαγάγουμε δεν μπορούν να είναι ε, μερικά, στρεβλωμένα και ακόμη μεροληπτικά. Γι' αυτό θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει με ένα δίκτυ πάνω στον οποίο θα στηρίζονται όλες οι πολιτικές. Το ΑΕΠ υπάρχει ως αποδεδειγμένα καλός δείκτης για να προσμετρηθεί ένα σύνολο πολιτικών. Έχει προσφέρει δηλαδή καλές γνώσεις των εξελίξεων, έχει επιτρέψει καλές επιλογές. Αλλά ο δείκτης του ΑΕΠ είναι ως εκ της ίδιας της φύσεως περιορισμένος ο πεδίο που μπορεί να καταγράψει. Δεν επιτρέπει δηλαδή την καταγραφή της προόδου, της ευημερία του ανθρώπου. Ε, δεν μπορεί το πόσο καλά αισθάνεται κανείς και το πόσο καλά ζει η ποιότητα ζωής του να υπολογιστεί με μια τέτοια οικονομική ε, καμπύλη. Έτσι λοιπόν τέτοιου είδους δείκτες στηριγμένοι αποκλειστικά στο ΑΕΠ ε, στρεβλώνουν την πραγματικότητα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, δεν την καταγράφουν επιστά και δεν επιτρέπουν ως εκ τούτου την αξιολόγηση της ε, ανθρώπινης ε, προόδου. Το ΑΕΠ μόνο του δεν μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο μιας πηξίδας να μας καθοδηγήσει δηλαδή και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω ε, περιπτωσιολογικά κάποιες άλλες ε, λύσεις όπως ανεργία, ε, κίνδυνος φτώχειας, υγεία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ποιότητα πλαισίου ζωής, ευημερία, ποιότητα πόρων, ποιότητα υδάτων και αέρος, πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, διάφορες μορφές ρήπανσης και ούτω καθεξής. Αυτά περιπτωσιολογικά μόνο. Και θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι συχνά, από την πρόσφατη ιστορία το διδασκόμαστε αυτό, υπάρχει ε, ρήξη μεταξύ της οικονομικής ε, προόδου και ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης, ε, την οποία καταγράφει κατά τρόπο εσφαλμένο το ΑΕΠ. Και γι' αυτό θέλουμε πέραν του ΑΕΠ να, ε, να συμπεριλάβουμε και έναν δείκτη ο οποίος θα καταγράφει τις πιέσεις βάρος του περιβάλλοντος, της ποιότητας περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής μας, δηλαδή της ε, ευημερίας μας τελικά. Και δεύτερον ένα δείκτη της ζωής και της ευημερίας που θα στηρίζεται σε κοινωνικούς, σε κοινωνικές ενδείξεις. Εάν λοιπόν θέλουμε μία πιο ολοκληρωμένη, πληρέστερη και αποτελεσματική ε, θεώρηση της περιφερειακής μας πολιτικής, πρέπει να έχουμε κατάλληλα μέτρα υπολογισμού και μέτρησης με κριτήρια τα οποία θα συμπληρώνουν το ΑΕΠ και που θα επιτρέπουν στην περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχής, να είναι πιο ορθολογική, να έχει καλύτερο τρόπο ε, εξέτασης των συνθήκων που επικρατούν σε διάφορες περιφέρειες, χάρη στους δείκτες αυτούς, να έχει καλύτερη αντίληψη και αντιμετώπιση ή ταξινόμηση τελικά των περιφερειών ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα ως προς την χρήση αυτών των νέων δικτών δεν υπάρχουν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης η πραγματική, η ουσιαστική θέση εφαρμογή μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαρκούς ανάπτυξης, η οποία σας υπενθυμίζω αγαπητοί συναδελφοί αποτελεί την ε, σπονδυλική στήλη, την ράχο κοκαλιά της ανάπτυξης και που ε, εκφράζεται κατά τρόπο συμπαγή από τις τρεις ε, συνιστώσεις της, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα κύριε Πρόεδρος. Ο Μιχαήλ έχει ζητήσει τον λόγο πρώτος. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είπε και ο συνάδελφος Μπεσέ μόλις τώρα ότι το ΑΕΠ είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε από καιρό εισαγάγει και αξιοποιούμε αποτελεσματικά για τον υπολογισμό της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, έχει ωστόσο ε, υποστεί επικρίσεις ως ε, δείκτης μέτρησης εδώ και αρκετό καιρό. Επικρίσεις οποίες έχουμε και εμείς συζητήσει στην Επιτροπή μας διεξοδικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε μια πολιτική συζήτηση για το, για το ΑΕΠ δεν μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα πολιτικά. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν, αλλά δεν ε, μπορώ να είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα έχουμε ικανοποιητική ε, προσμέτρηση των δεδομένων με κάποιους άλλους δείκτες, πρόσθετους δείκτες. Και θα ήθελα εδώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το εξής. Καταρχάς να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η ιδέα που θα έχουμε του κατά πόσο είναι μετρήσιμοι αυτοί οι δείκτες, πραγματικά μετρήσιμοι, και επίσης το κατά πόσο αυτοί οι δείκτες είναι εκτεθειμένοι σε αξιολογικές κρίσεις. Τι σημαίνει ευημερία, τι σημαίνει ευτυχία. φαίνεται ότι με το εισόδημα ή με τις οικονομικές ε, μεταφορές οικονομικών ε, ε, στοιχείων δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κανείς εξασφαλίσει την ευτυχία ή όχι. Δεν είναι δεδομένοι δηλαδή οι συσχετισμοί μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και των παραγόντων όπως η ευημερία ή η αίσθηση της ευτυχίας. Άρα όταν είναι να κάνουμε συγκρίσεις ή υπολογισμούς θα πρέπει αυτούς τους υπολογισμούς και αυτές τις συγκρίσεις να τους κάνουμε με ίσα πράγματα, δηλαδή αν είναι να μιλούμε για, οικονομικά, για οικονομικές αξίες, να τις υπολογίσουμε με οικονομικούς δείκτες και ούτω καθεξής γιατί και εγώ που έχω να παρελθόν ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους δείκτες. Είχαμε παραδείγματι την εισαγωγή στο Βάδι Βιτεμβέργη τέτοιου είδους νέων δικτών στην ε, περιοχή μας, εθνικών δικτών, όπου όμως κατέστη καθοριστική σημασίας το πόσο πόση ανάπτυξη θέσεων εργασία είχαμε, όχι το πόσε θέσει εργασία σε απόλυτο αριθμό. Και άρα μια περιοχή, μια περιφέρεια ή ένα κομμάτι περιφέρειας το οποίο είχε μια ικανοποιητική ανάπτυξη ήταν αυτό που είχε αρκετή αύξηση θέσεων εργασίας. Ενώ μια άλλη που φαινόταν ότι έχει καλή οικονομική ανάπτυξη είχε μια, παρουσίαζε στασιμότητα ως προς τη δημιουργία των θέσεων εργασίας. Άρα εδώ έχουμε να κοιτάξουμε περισσότερο την δυναμική, την εξέλιξη δηλαδή και όχι την στατική εικόνα που παρουσιάζει μια περιφέρεια. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί κανεί να θεωρήσει ω ελκυστική λύση, δηλαδή την εισαγωγή διαφορών δικτών τα λοιπά και μπορεί να υπάρχει και σχετική φιλολογία. Εγώ όμω βλέπω και από την πρακτική μου και από την εμπειρία μου δηλαδή ότι αντιμετωπίζουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή ότι αυτό ο παλαιό δείκτη, ο οποίο έχει αποδείξει τι αδυναμίε του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα νέο δείκτη, ο οποίο ναι μπορεί να τον συμπληρώνει, αλλά αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι δεν είναι ε, αρκετά καλά μελετημένος και σχεδιασμένος και πάνω απ' όλα δεν την χάνει συνένεση. Άρα καλοί οι δείκτες, αλλά θα ήθελα επαρκή ενημέρωση, επαρκή τεκμηρίωση, επιστημονική συζήτηση και να γνωρίζουμε στα τελευταία ανάλυση τι είναι αυτοί οι δείκτες, να το έχουμε προκαθορίσει πριν από την εισαγωγή τους και να ε, συζητήσουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας όσο το δυνατόν εντατικά το ζήτημα αυτών των δικτών. Να ζητήσουμε να έρθουν ενδεχομένω και εμπειρογνώμονε, να συστήσουμε μαζί του τα θέματα των δικτών πριν καταλήξουμε στην λήψη μια αποφάσεω για τη συμπλήρωση του δίκτυ. ΑΕΠ με κάποιου άλλου δείκτε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουσάνα Προσφόχα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την αυτή πρόταση, τη μελέτησα. Εάν χρησιμοποιήσουμε περισσότερους δείκτες, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Πρέπει βέβαια πρώτα να εντοπίσουμε τους δείκτες και να ε, έχουμε και μια καλή εικόνα της μεθόδου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την κατάρτιση των δικτών αυτών, πώς θα τους καταρτίζουμε, πώς θα τους υπολογίζουμε, με ποιες παραμέτρους. Για το περιβάλλον, Φερρυπίν, υπάρχουν παράμετροι που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μέσα σε διάφορα σχέδια, project κτλ. Project τα οποία ασχολούνται με την ποιότητα των υδάτων ή του αέρος. Παράμετροι οι οποίες όμως σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, όπως για παραδείγμα στην απασχόληση ή την εκπαίδευση. Μπορούμε λοιπόν τέτοιου είδου, είδους ε, δείκτες να τους χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε ενδεχομένως την εικόνα που έχουμε, τη γνώση που έχουμε για μια περιοχή, μια περιφέρεια, αλλά μπορούμε τους είδους αυτούς δείκτες να τους χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε κάποια μέτρα, να έχουμε καλύτερα μέτρα πολιτική. Ο δείκτης της ανεργίας, Φερρυπίν. Ο δείκτης της εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία. Πώς καταγράφονται οι άνεργοι στην κάθε χώρα. Ποιος μπαίνει μέσα στις στατιστικές αυτές. Και για πόσο καιρό μένει μέσα. Επομένως, καθώς τα συστήματα διαφέρουν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αξιόπιστο σύστημα καταγραφής της δείκτη. Επίσης, ευτυχία η ευημερία. Πώς, πώς την υπολογίζουμε. Μπορούμε φερειπή να συμφωνήσουμε όλοι ότι μία μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Πολύ καλά. Αλλά μπορεί να ε, ανησυχούν οι περίοικοι ότι οι δυσάρεστοι σωσμές θα επιδεινώσουν την ποιότητα, θα επιβαρύνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος τους. Ε, τέτοια και άλλες παράμετροι μπορεί να επισημάνουν αντίστοιχα προβλήματα. Έχουμε ήδη λάβει την απόφαση που θα μας επέτρεπε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα διαρθρωτικά ταμεία. Εάν όμως αγάγουμε περισσότερες παραμέτρους και δείκτες, η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα δεσχεράνε, θα περιπλακεί. Και γι' αυτό εγώ προτιμώ πάντοτε να είναι απλές οι παράμετροι ή οι δείκτες που χρησιμοποιούμε, εύκολα μετρήσιμοι. Και πάντοτε οι δείκτες να είναι σχετικοί με το θέμα ή το project για, τον οποίο, για το οποίο χρησιμοποιούνται. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ο κύριος Πίπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Τόιρερ ότι θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε μία ακρόαση για το θέμα αυτό του δίκτυου του ΑΕΠ. Συστήθηκε άλλωστε και χθε από τους συντονιστές το ίδιο θέμα. Είναι καλή ιδέα πιστεύω. Εμένα πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιδέα δεν μου κινεί επουδενή το ενδιαφέρον. Είναι μία προσπάθεια των πρασίνων οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με διάφορες πτυχές του Κοινοβουλίου. Μια προσπάθεια λοιπόν να ανατρέψουν μια αξιόλογη και αποδεδειγμένη αξιόλογη ε, μονάδα μέτρησης που έχουμε και αυτό μόνο για ιδεολογικούς λόγους, το ΑΕΠ δηλαδή. Είναι μια σαφής προσπάθεια η οποία πάντως θα σήμαινε ταυτόχρονα και τη διάλυση, διάλυση της αλληλέγγυας ε, κοινωνίας που έχουμε ε, χτίσει εδώ οικονομίες στην Ευρώπη, διότι εάν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, εάν επιτρέψουμε την παρισύφρηση ε, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων δικτών σε ίσους όρους με αυτούς του ΑΕΠ, ουσιαστικά κηρύσουμε τη διάλυση της αλληλέγγυας δικαιοσύνη, κοινωνίας ε, όπως σε παραδείγματι εμείς στη Γερμανία που έχουμε ε, σε ορισμένες περιοχές μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περιοχή που είναι εγκατεστημένη η Μπάσφε, παραδείγματι, η χημική βιομηχανία στη Γερμανία, που είναι ευημερούσα αλλά με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό θα οδηγούσε λοιπόν σε ανατροπή κάθε είδους ε, αξίας και προγράμματος που έχουμε και μάλιστα θα άνοιγε πορτοπαράθυρα με εισαγωγή τέτοιων δικτών στην αυθαιρεσία. Επομένως προβλήματα όπως η ανεργία, οι κλιματολογικές αλλαγές, ειδικά προβλήματα περιβαλλοντικής ρήπανσης ή του περιβάλλοντος. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κατά τρόπο ευφύη, με ευφύη αξιοποίηση των στατιστικών που έχουμε στη θέσή μας κατάλληλη αξιοποίηση των στατιστικών, αλλά όχι έτσι. Μια περιοχή η οποία είναι φτωχή, που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του ΑΕΠ, δεν είναι σε θέση βέβαια να κάνει καμία επιπλέον προσπάθεια ή δαπάνη υπέρ του περιβάλλοντος. Γι' αυτό έχουμε την πολιτική της συνοχής και γι' αυτό θέλουμε να τη συνδυάσουμε με την πολιτική της Ευρώπης του 2020, με κοινωνική πολιτική, με περιβαλλοντική πολιτική ενσωματωμένη, οι οποίες θα αποβούν εις των πιο φτωχών προβλημάτων, θα του επιτρέψουν και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά του προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλλά όχι τώρα να ανατρέψουμε έναν δείκτη μόνο και μόνο γιατί οι πράσινοι θέλουν για να ικανοποιήσουν την πελατεία του τι μη κυβερνητικέ του οργανώσει και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διασφαλίσουν την επικράτησή του με τι νέε ε, αποκεντρωμένε υπηρεσίε που έχουν εξασφαλίσει ε, και να ικανοποιήσουν μόνο αυτή τους την πολιτική. Εδώ πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα και να πούμε όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και εμεί ω περιφερειακή πολιτική, γιατί δεν είμαστε η Επιτροπή του Περιβάλλοντο, πρέπει να πούμε ένα ξεκάθαρο όχι. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Τυρολιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Η έκθεσή του, το έγγραφο αυτό που συνέταξε, νομίζω θα μας δώσουν ιδέες για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τα ζητήματα αυτά που μας ενδιαφέρουν και το πρόβλημα του ΑΕΠ με τους δείκτες του. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο όλο ζήτημα των δικτών ανάπτυξης και για σκοπούς συλλογική εξέλιξης θα πρέπει να κάνουμε τους δείκτες αυτούς όσο πιο εύχριστους και να λαμβάνουμε όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα της επικυροποίησης των ολοκανόνων από την πλευρά της Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή είναι ένα κείμενο για να εξισορροπήσουμε και πάλι τις καταστάσεις, για να δώσουμε μια θέση πιο σημαντική στον προβληματισμό τον περιβαλλοντικό που θεωρούμε πολύ ε, σημαντικό του. Είναι λοιπόν ε, σκόπιμο όλα αυτά. Απλώς το κείμενο θα ήταν πιο εύστοχο εάν παρουσίαζε την κατάσταση και των οικονομικών δικτών ε, συνοψίζοντας και τους εναλλακτικούς δείκτες που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να δοθεί ως πρόταση του εισηγητή και ενώ προσυπογράφω γενικώ τις προτάσεις του, νομίζω ότι δεν είναι απλό για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού να προβλέπουμε αξιολόγηση των ε, περιοχών βάσει των δικτών τους. Επίσης, πιστεύω ότι για να είναι αποτελεσματική η περιφερειακή πολιτική και στον ε, τομέα του περιβάλλοντος, της πρόσβασης της τεχνολογίας της πληροφορίας, ε, την ε, απασχόληση θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης για την πολιτική συνοχής με σημαντικούς δείκτες προτεραιότητας. Ευχαριστούμε κυρία Σρέτερ. Νομίζω θα πρέπει εδώ να διασκεδάσω κάποιους μύθους. GDP Beyond, πέραν του ΑΕΠ δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν ξεκίνησαν οι πράσινοι, αλλά ο Σαρκοζή ο ίδιος στον ΩΣΑ και μάλιστα τον επικρότησαν πολύ και εμείς βεβαίως, αλλά σας διαβεβαίω ότι ο Σαρκοζή δεν είναι μέλος των πρασίνων, ούτε καν του, του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Επίσης, στην, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η κύρια ομάδα, η μεγαλύτερη ομάδα είναι το ΕΛΚΑ και έχει τη σχετική έκθεση από την ομάδα των, πώς το λένε αυτούς, την ΕΕΔΕ τους, ε, της Ευρώπης των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών. Δεν θυμάμαι πώς το λέμε αυτό στα γερμανικά. Η συγγήτρια για τη γνωμοδότηση στην κοινωνική πολιτική, στην κοινωνική επιτροπή είναι η κυρία Χάρτλινγκ, που δεν είναι πάλι από τους πρασίνους, αλλά από τους φιλελεύθερους βουλευτής. Και το θέμα αυτό εμείς το θεωρούμε και σημαντικό και σκόπιμο, σωστό. Όπως υπόθηκε δηλαδή, το ΑΕΠ αποδεικνύεται ότι δίνει μόνο στρεβλωμένη και μονοδιάστατη εικόνα της κατάστασης. Στο πρώτο αυτό δε έγγραφο εργασίας μιλούμε μόνο για την εισαγωγή ε, πρόσθετων δικτών και όχι για κατάργηση του ΑΕΠ. Δικτών δηλαδή οι οποίοι απλώς θα αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπου δεν είναι σαφής η εικόνα. Να σας ένα παράδειγμα. Ξέρουμε πολύ καλά τι υπολογίζεται με το ΑΕΠ ε, και ότι το ΑΕΠ ας πούμε καταγράφει και επενδύσεις, χρήμα που ε, εισραίει σε μια περιφέρεια. Μια φτωχή περιφέρεια η οποία ε, εισπράττει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπει την αύξηση του ΑΕΠ της αυτομάτως, χωρίς όμως να εξετάζεται εάν με τις επενδύσεις αυτές, με τις επιχορηγήσεις αυτές δημιουργούνται νέες εργασίας, εάν βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, εάν είναι καλύτερη η κατανομή του εισοδήματος. Δεν είναι λοιπόν αυτόματη η βελτίωση της κατάστασης σε μιας περιοχής. Ενώ ο δείκτης του ΑΕΠ αυτό κάνει. Με το που εισραίουν τα χρήματα στην περιφέρεια αμέσως αυξάνεται και δίνει διαφορετική και στρεβλωμένη εικόνα. Αυτό το αποδεικνύουν σε τελευταία ανάλυση και πολλές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν εντοπίσει το πρόβλημα από το 2000 ήδη. Ε, πολλές πραγματικά μελέτες οι οποίες επισημαίνουν το πρόβλημα και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να εξετάσουμε εάν το ΑΕΠ είναι το άπαν και αν χρειάζεται να εισρέψουν και άλλα κριτήρια στο σύστημα που θα χρησιμοποιούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένες ιδέες δεν ε, θα πρέπει να συζητηθούν. Αλλά εδώ ε, αυτό που θέλουμε είναι μόνο διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες ή μελέτες, στατιστικές αν θέλετε, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο κράτος και μπορούν σε διεθνές επίπεδο να ε, χρησιμοποιηθούν. Είναι ένα κριτήριο αυτό για την επιλογή ενός δεκτήτου, να είναι, το να είναι δηλαδή διεθνώς αναγνωρισμένος, να χρησιμοποιείται από κάποιο κράτος μέλος με τρόπο αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει ζήτημα δηλαδή να πούμε ότι εισάγουμε κάποιον δίκτυο ο οποίος δεν είναι αποδεδειγμένα αποδεδειγμένα ε, σε κάποιο κράτος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δείκτες που προτείνουμε, οι οποίοι υπάρχουν, χρησιμοποιούνται και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα ή νέους δείκτες, αλλά να αξιοποιήσουμε αυτούς που ήδη υπάρχουν. Ε, πρέπει να πω ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ ισορροπημένη, είναι εμπεριστατωμένη και ταυτόχρονα επισημαίνει ξεκάθαρα τα σημεία στα οποία χρειαζόμαστε βελτίωση έτσι ώστε να μην μένει μια περιοχή ε, ως τελευταίος τρεχός της στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το ΑΕΠ καταγράφοντα μόνο ένα, ε, μία όψη της κατάστασης δεν μπορεί να δει τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να έχει αυτή η περιοχή. Γι' αυτό θέλουμε τα, τα χρήματα που δαπανούμε και με προγράμματα όπως το Τζίνι και άλλα να ε, αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Κατά τα άλλα, το έργο εργασία του εισηγητού, του συντάκτη, είναι πάρα πολύ καλό και αποτελεί μια συμβολή, μια παρέμβαση στη συζήτηση. Θα ήταν βέβαια και παράλογο η Περιφερειακή Επιτροπή να μην γνωμοδοτήσει στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Αλφόνση. Ο κύριος ε, Αλφόνση. Πρώτα απ' όλα να πω στον συνάδελφο Πίπερ ότι μας ε, επικρίνει για την ιδεολογική μας προσέγγιση, όμως βρίσκω ότι και εκεί η δική του παρέμβαση γεμάτη από ιδεολογικά στοιχεία ήταν. Σε κάθε περίπτωση για το ζήτημα αυτό, όπως είπε και η Μπεθ, είναι αυτό ένα στοιχείο για το οποίο ανησυχούν όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι πράσινοι. Και είναι και επίκαιρο το όλο ζήτημα, διότι θα περάσουμε σε μια νέα περίοδο προγραμματισμού. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ερωτήματα για το κατά πόσον είναι αρκετά τα κριτήρια του ΑΕΠ και μόνον αυτά δεν λέω να μην εξετάσουμε τις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και με τα στοιχεία του ΑΕΠ, αλλά θα πρέπει σαφώς να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Ένα κοινωνικό κριτήριο που μου φαίνεται αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το κόστος του, της ζωής. Ε, σε χώρες, σε περιοχές όπου έχουν ε, λόγω χάρη μεταξύ τους ίσο ΑΕΠ, αλλά πολύ διαφορετικό κόστος ζωής, ε, προφανώ οι πληθυσμοί δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν ε, είναι ισότιμε οι συνθήκε διαβίωση. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί λοιπόν υπόψη. Επίση, περιβαλλοντικά κριτήρια. Αναζητούμε το πώ θα προβάλλουμε ευρωπαϊκέ πολιτικές με και οθυλή συμμετοχή των πολιτών, λόγω χάρη για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό το κριτήριο λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στην επιλογή του στήριξη που θα παρέχουμε στην περιφερειακή πολιτική. Ένα παράδειγμα. Βρίσκομαι σε ένα νησί, ας πούμε. Υπάρχουν δύο προγράμματα για οικοδόμηση λιμένος ε, ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ένα που το στηρίζει η βασική πόλη στην οποία θα χτιστεί το λιμάνι και ένα από μια μικρότερη πόλη. Ε, αλλά τι είναι το σημαντικό, ε, ότι αν χτιστεί το λιμάνι αυτό θα ε, περιοριστεί η απόσταση μετροπολιτικής Γαλλίας και Κορσικής κατά τρεις ώρες, ε, τρεις ώρες θα κρατάει το ταξίδι οπότε θα μειωθεί και η εκπομπή ε, διοξιδίου του άνθρακα με τη μείωση αυτή του χρόνου του ταξιδιού. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει τέτοιο είδους μέρημνα όταν επιλέγουμε τα προγράμματα και ποια θα στηριχτούν, να είναι περιβαλλοντικό κριτήριο. Μα ζητάτε λοιπόν τώρα να μελετήσουμε με τρόπο μάλλον αντικειμενικό και όχι με ιδεολογικές προκαταλήψεις. Η κυρία Κρέλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ενδιαφέρον είναι το ότι συνεχίζω στα όσα μόλις υπόθηκαν. Μια, μια προκατακτική μάλλον παρατήρηση. Πριν από ένα χρόνο περίπου, συνομιλώντα με έναν συντονιστέ για το αν θα μπορούσαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή να συμφωνήσουμε το να είναι στο να είναι η Περιφερειακή Επιτροπή ε, κατ' ουσίαν αρμόδια, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είχα αναγνωρίσει τη μεγάλη σημασία της ε, υπόθεσης αυτής, δηλαδή δεν επέμεινα όσο θα έπρεπε για να είναι η Περιφερειακή Πολιτική Επιτροπή κατ' ουσίαν αρμόδια, ενώ θα έπρεπε πιστεύω τώρα πια, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Για την Περιφερειακή Πολιτική, την πολιτική συνοχή, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, σχέδια, όπου χωρίς δυσκολία θα μπορούμε δείκτες άλλους από το ΟΑΕΠ να τους εισάγουμε, να τους χρησιμοποιούμε και αυτό πιστεύω ότι ακόμη και από την οπτική γωνία του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος μπορεί να είναι ενδιαφέρον και μπορεί να εισαγόνται και, άλλες, και άλλα θέματα προς συζήτηση, αλλά πάντως εμείς ως περιφερειακή πολιτική πρέπει εξάπαντος να επιμείνουμε στην εισαγωγή της πολιτικής της συνοχής μέσα στην ε, προσμέτρηση αυτή και έχουμε δαπανίσει αρκετό χρόνο και να συζητούμε την πολιτική συνοχής με τροπολογία στην οποία καθιστούμε σαφές ότι το ΑΕΠ παραμένει κύριο κριτήριο για τον υπολογισμό της ε, για την, πολιτική της, ε, την περιφερειακή πολιτική και συμπληρώνεται από άλλους δείκτες εφόσον αυτοί έχουν αποδεδειγμένα κριθεί ικανοποιητική όπως υπόθηκε και νωρίτερα, αλλά επιμένουμε ότι παραμένουμε με κύριο δείκτη το, το ΑΕΠ. Ε, για δεν την προηγούμενη μόλις παρέμβαση, θα ήθελα να πω ότι σχεδόν με αναγκάζει να πω ότι το κόστος ζωής, το κόστος διαβίωσης, σημαίνει ότι μεγαλύτερες πόλεις όπως το Μόναχο που έχουν το υψηλότερο κόστος ζωής στη Γερμανία Φερρυπίν θα χρειάζονται και ενίσχυση διότι είναι τόσο υψηλό το επίπεδο διαβίωσης, τόσο υψηλό το κόστος μάλλον ζωής που θα χρειάζονται βοήθεια <coughs> οι άνθρωποι. Ε, είναι παράλογο αυτό. Όχι. Το κόστος ζωής είναι βέβαια θέμα προσυζήτηση αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και δείκτες οι οποίοι δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε τυχαία να βρίσκουμε ένα κριτήριο ή ένα θέμα και να λέμε «Α, αυτό θα είναι δείκτης». Γιατί δεν μπορούμε τότε να έχουμε προσμέτρηση και υπολογισμό ε, σε όλη την Ευρώπη κατά τρόπο ισότιμο και ισοδύναμο και εδώ ακριβώς το σχέδιο για το project αυτό για τα λιμάνια δείχνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση ενδεχομένως σε μια περιοχή συγκεκριμένη να βλέπουμε κάποια ε, διαφορετικά κριτήρια αλλά αν θέλουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε ποιος χρειάζεται υποστήριξη, ποιος χρειάζεται ενίσχυση μέσα από την πολιτική της συνοχής μόνο το ΑΕΠ μπορούμε να έχουμε ως δείκτη και εάν είναι δυνατόν, εάν χρειάζεται δείκτες μετρήσιμους που όμως είναι μετρήσιμοι με βάση τους ίδιους ακριβώς στατιστικούς κανόνες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ε, ακολουθούν τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις. Να σας πω, εγώ από την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ε, θυμάμαι μία φράση ε, για το τι είναι ο στατιστικολόγος. Ο στατιστικολόγος είναι αυτός ο οποίος πειράζει τα στατιστικά στοιχεία. Ε, δεν θέλω βέβαια να κατηγορήσω τη Eurostat για τίποτε τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αν εφετέρου δεχόμαστε δείκτες που θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και θα οδηγούν σε κατηγοριοποίηση στοιχείων όπως φτώχεια, βημερία ε, και ούτω καθεξής, χωρίς ε, να τους μελετήσουμε και να τους διευκρινίσουμε περισσότερο τους δείκτες αυτούς. Γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στην εισαγωγή νέων δικτών. Εάν παραδείγματι υποθεί ότι να νέα στατιστικά στοιχεία ε, που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ. Φέρει πίν, ανεργία που όλοι επισημαίνουν. Ναι, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την ανεργία ως δείκτη, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται είναι πάντοτε η ίδια και παντού. Ε, και επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε και υπόψη ότι χρειάζεται περιορισμό της γραφειοκρατίας φερρυπίνος ιδεώδες. Μήπως θα πρέπει να έχουμε και άλλους δείκτες ε, για το πόσο ορατή είναι η Ευρώπη, πόσο ανοιχτή είναι μια περιφέρεια στην εξέλιξη κτλ. Ε, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σε περιφερειακό επίπεδο δεν θα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε, ή δείκτε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα επιβάλλουμε εμεί ω Ευρώπη, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εάν θέλουν μέσα σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια διαφορετικού δείκτε από τα κράτη-μέλη, τότε οφείλουν να το πράξουν τα κράτη-μέλη αυτό. Εμεί θα πρέπει να είμαστε σε θέση με του δείκτε που θα έχουμε του Ευρωπαϊκού, να βλέπουμε αν κάποια περιοχή έχει περισσότερη ανάγκη για υποστήριξη, εάν χρειάζεται να ενταχθεί στην πολιτική συνοχή κ.ο.κ. Ευχαριστώ κύριο Σούλτνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, εξ ονόματος του ΕΛΚ, και ως ασκαιώδης εισηγητής της ομάδας αυτής, να πω ότι πρέπει να είμαστε βεβαίως ανοιχτόμυαλοι στην προσεγγίση μας εδώ. Οι διάφοροι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο πρόσφορο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς στην επιλογή μας. Για την ώρα δεν έχουμε βεβαίως άλλους δείκτες πέραν του ΑΕΠ δείκτες στους οποίους να μπορούμε να βασιστούμε για να κατανείμουμε τις διάφορες μορφές βοήθειας, υποστήριξη προς τις επαρχίες και τις περιοχές της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκπονηθούν διαφορετικές μελέτες ή ότι δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ε, παραδείγματα κακής υλοποίησης όπως και πάρα πολύ καλής. Και σίγουρα οι δείκτε του ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο τη διαβίωση των πολιτών, όμω για την ώρα δεν έχουμε τίποτε καλύτερο και τίποτε πιο αυθεντικό στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε. Έχει αποδειχθεί και μάλιστα εδώ και χρόνια ότι το, ε, η εσωτερική κατανομή των δικτών του ΑΕΠ θα μπορούσαν να εξεταστούν και να αναδιορθωθούν. Όμως το εργαλείο αυτό είναι σαφώς χρήσιμο. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι η αλλαγή των δικτών θα αντικατοπτρίζει και διαφορετικές καταστάσεις. Σίγουρα διαφορετικές μέρημνες πρέπει να καλύπτονται από τους δείκτες, αλλά και σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης είναι σκόπιμο να βεβαιωθούμε ότι θα είναι αποτελεσματικά αυτά που θα προβλέψουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η απόφαση που ελήφθη μέσω της ψηφοφορίας ήταν ε, ορθή, διότι από τη μια ανοίγουμε την ε, προσελκύουμε μάλλον το ενδιαφέρον και έπειτα ε, τονίζουμε ότι πρέπει η κατανομή να γίνει προσεκτικά. Να λάβουμε υπόψη το τοπικό ΑΕΠ. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι μεταξύ κρατών, περιοχών, περιφερειών. Θα πρέπει εδώ να υπάρξει monitoring, παρακολούθηση. Διότι εξ εμπειρίας γνωρίζουμε ότι κάποιοι δείκτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ακόμη και σε επίπεδο ένωσης. Στη φάση όμως που βρισκόμαστε τώρα, απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ η γνωμοδότηση που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή να περιέχει υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Αυτή είναι η γενική άποψη του ΕΛΚ. Η, έκθεσή μας θα πρέπει να επιτρέψει την εισαγωγή καινοτομιών. Σίγουρα περιέχει κάποιες ωραίες φράσεις γιατί με τη σημασία του ΑΕΠ, το κείμενο που λάβαμε, όμως Φαίνεται εδώ να υπάρχουν ευγενικέ διπλωματικέ διατυπώσει και όχι ουσία. Ίσως υπάρχουν και διαφορετικές ευαισθησίε στον τομέα αυτό, αλλά είναι καθησυχαστικό να βλέπουμε ότι κατά τη συζήτηση για το θέμα αυτό δεν υπάρχει σοβαρή απόκληση μεταξύ των εκπροσώπων των νέων και των παλιών κρατών μελών. Υπάρχουν περισσότερο προσωπικές τοποθετήσεις. Τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλωστε είναι αυτά που κατεξοχήν στο, στηρίζουν την επιλογή του ΑΕΠ ως του προτιμόμενου δίκτυ. Άρα το ΕΛΚ θεωρεί ότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας θα πρέπει να τροποποιηθεί. Επί της ουσίας. και επειδή Έχω ακούσει προσεκτικά τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιφέρουμε τώρα σημαντικέ αλλαγέ. Φυσικά, να εξετάσουμε ποιοι θα είναι οι δείκτε προτεραιότητα που θα χρησιμοποιήσουμε μετά το 2004. Όμω προ στιγμή εκφράζουμε απλώ απόψει. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε την κατάληξη τη συζήτηση. Βεβαίω τα πράγματα θα εξελιχθούν. Όμως, για να παραμείνουμε στο παρόν, επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι ακόμη. Να, να θυμίσω μία έκφραση. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από την πεπατημένη. Εάν είμαστε βέβαιοι για τη νέα μας επιλογή, αν θέλουμε να λοξοδρομήσουμε, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι παίρνουμε τη σωστή κατεύθυνση, τότε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να είναι περιστατωμένη αυτή η επιλογή. Όπως όταν αλλάζει, ο εκλογικός νόμος σε ένα κράτος μέλος. Ξέρουμε ότι ε, λόγω της αλλαγής μπορεί να αλλάξει και η μορφή της εντολής που έχει ο ένας ή ο άλλος φορέας και επίσης η κατεύθυνση της προφορίας των του εκλογικού σώματος. Εδώ λοιπόν η πρόταση αυτή είτε προέρχεται από την Επιτροπή είτε τε από το Κοινοβούλιο, εφόσον επιφέρει αλλαγή, πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Πρέπει να δούμε μήπως επηρεαστεί σοβαρά η πολιτική συνοχή. Οι μελέτες που εγώ γνωρίζω και έχω υπόψη μου δεν κάνουν προτάσεις ιδιαίτερα ριζοσπαστικές. Πρέπει να παραμείνουμε στα γνωστά πλαίσια. Καλές είναι οι νέες λύσεις, καλό είναι να προσέχουμε τις εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου, όμως Δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν πρέπει να πάμε πολύ μακριά. Η Κορσική άλλωστε, για να έρθω και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν είναι μια εξόχως απομακρυσμένη περιοχή. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από άλλες περιοχές. Από μια μη νησιωτική περιοχή, όμως για την ώρα φαινόταν να υπάρχει ένα σύστημα που ευνοεί περιοχές της περιφέρειας που βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση από ό,τι άλλες. Όπου οι δείκτες δεν επαρκούν για να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα των δυσκολιών τους. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να μην επιμένουμε στην αλλαγή για την αλλαγή των δικτών. Πρέπει λοιπόν να δούμε που υπάρχουν υψηλοί δείκτες, αλλά και που χαμηλότεροι. Και για όσους είναι πράσινοι στο πνεύμα, θα πρέπει να μην ξεχνούν ότι σημαντικό είναι πώς τελικά θα εκτελεστούν τα κονδύλια δάση των δικτών του ΑΕΠ. Είναι πολύ καλό το παράδειγμα της Κορσικής, και αν επενδύσει συγκεκριμένε είναι πιο ωφέλιμε για το περιβάλλον, σαφώ πρέπει να προτιμηθούν από άλλε που θα είναι βλαβερέ για το περιβάλλον. Είναι προφανέ αυτό. Όμω, μια συγκεκριμένη, μια δεδομένη περιοχή θα πρέπει να δούμε αν χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη στήριξη βάσει του γενικότερου πλαισίου. Έπειτα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα προγράμματα, το υπάρχον πλαίσιο πρέπει να αξιοποιείται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Θα πρέπει σίγουρα εδώ να μας οδηγούν και οι οικολογικές μέρημνες. Όμως οι πολιτικές ομάδες πιστεύω ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν για κοινό σκοπό αλλά δεν μπορούμε και να παραβλέπουμε τους υπάρχοντες δείκτες. Δείκτες που είναι δοκιμασμένοι στο χρόνο, δείκτες που κατανέμουν την στήριξη μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων περιοχών τους. Να πως ε, αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Οι τροπολογίες μας θα έρθουν εν ευθέτω χρόνο μαζί με των υπολείπων πολιτικών ομάδων. Ευχαριστούμε κύριο Σωρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα να σας πω ότι κανείς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος στα προβλήματα που φύγει ο εισηγητής μας. Άλλωστε το αποδεικνύει αυτό και η συζήτηση που κάναμε μόλις. Εδώ μου φάνηκε να αντιλαμβάνομαι από τα λόγια κάποιων συναδέλφων, του εισηγητή μάλλον, ότι δεν προτείνει την κατάργηση των δικτών του ΑΕΠ, θεωρεί ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, αλλά που είναι κάπως περιοριστικό για να καταμετρά την πρόοδο μιας ολόκληρης κοινωνίας και θεωρεί ότι καλό θα ήταν πέραν του ΑΕΠ να εξεύρουμε και άλλα εργαλεία. Δεν λέω ότι τα πράγματα, ότι κάτι τέτοιο είναι απλό ω προσπάθεια, Όμω να πω στου συναδέλφου ότι ήδη η Ευρώπη στην πολιτική συνοχή τη θεωρεί ότι το ΑΕΠ δεν είναι το μόνο κριτήριο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Περιοχές που είναι επιλέξιμες για τον στόχο 1 των διευθυντικών ταμείων. Για να είναι επιλέξιμη μια τέτοια περιοχή για το στόχο αυτό υπάρχουν βεβαίω οι δείκτε του ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε βεβαίως να κάνουμε την όλη συζήτηση αυτή, αλλά να είμαστε και ανοιχτόμυαλοι, διότι προφανώς μπορούμε να θεωρούμε ότι το ΑΕΠ καλό είναι να διατηρηθεί, σαφώς, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε με άλλα στοιχεία αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό καλό θα είναι να γίνει συζήτηση με εμπειρογνώμονες και νομίζω ότι είμαστε όλοι αρκετά ευφύς ώστε να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία. Σίγουρα δεν είναι απλό να δούμε από ποσοτικής άποψης το ένα ή το άλλο κριτήριο. Όμως ας έχουμε την τόλμη να ξεκινήσουμε αυτού του είδους την ανταλλαγή απόψεων ίσως θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα έτσι περαιτέρω. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και αν τα καταφέρουμε η Ευρώπη πραγματικά θα αποτελέσει υπόδειγμα και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα και για άλλες κοινωνικές ομάδες. Ε, ε, Ζεζίνα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Ως προς το στόχο που είναι η ενίσχυση των περιφερειών που έχουν καθυστερήσει σε σχέση με τις υπόλοιπες. Βεβαίως ε, το ΑΕΠ είναι ένας πολύ καλός δείκτης για τη σωστή κατανομή. Για να υπάρχει... Για να δούμε ποιες είναι οι περιφέρειες που ε, έχουν ε, καθυστερήσει και ποιες είναι πιο ανεξάρτητες ε, και κάπως πιο αυτάρκεις. Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε των κριτηρίων αυτών και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτόν τον δείκτη. Είναι κάπως παράδοξοι οι υπόλοιποι δείκτες, ε, όπως για παράδειγμα η ευημερία και η πιο ευχαριστημένοι πολίτες. Όμως οι πιο ευχαριστημένοι πολίτες μπορεί να είναι στις φτωχότερε περιοχές και πρέπει να δούμε πώς αυτές ε, οι περιοχές ε, ανταποκρίνονται και στα υπόλοιπα κριτήρια. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο δείκτης του ΑΕΠ μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση των ε, <coughs> ηλεκτροτικών ταμείων Ενδεχομένως όμως να μιλούμε μόνο για κάποιες ποσοστιαίες ε, μονάδες. Από ό,τι κατάλαβα, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετους δείκτες, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε μόνο για άκρος απομονωμένες περιοχές, για νησιωτικές περιοχές, ε, όπως είπε και ο κύριος Σέριαν. Αλλιώς ε, η πολιτική θα καταλήξει σε παράδοξο και θα αναστατωθεί το όλο σύστημα. Θα φτάσουμε στο παράλογο δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σκόπιμο να γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα και Νομίζω ότι σημαντικό θα είναι να οργανώσουμε και μια συζήτηση πιο ε, εμβαθυμένη για, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ειδικών. Σαφώς ε, το κριτήριο του ΑΕΠ θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο. Σαφώς είμαστε υπέρ του ΑΕΠ, αλλά όχι μόνον. Το ΑΕΠ αυτό καθεαυτό η χρήση του ΑΕΠ ως κριτηρίου δηλαδή δεν μας επιτρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν κοιτάξει κανείς το μέλλον, μα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλήρως τις μελλοντικές προκλήσεις βασιζόμενοι στο ΑΕΠ. Εγώ έρχομαι από την ε, Φιλανδία που είναι αραιοκατοικημένη. Και υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα ακριβώ λόγω τη αραιή τη κατοίκηση. Ε, λόγω χάρη προβλήματα αντιγωνιστικότητα. Δεν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τέτοιου είδου δείκτε ω προ την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται λοιπόν διασύνδεση μεταξύ των δικτών που θα χρησιμοποιηθούν και των στόχων της στρατηγικής του 2020. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι και πώς μπορεί να επηρεάζονται από την ανταγωνιστικότητα ή την οικονομία. Ε, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά ποιοι είναι οι περιφερειακοί δείκτες που θα μας επιτρέψουν να ε, επιζητήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξη των στόχων μας. Για τους περιβαλλοντικούς επίσης δείκτες νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικοί και στο μέλλον. Ήδη υπόθηκε και νωρίτερα ότι έχουμε τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε λόγω των δημογραφικών αλλαγών, ακόμη και από την άποψη του ανταγωνισμού. Ίσως χρειάζεται ένας δείκτης που να συσχετίζει λοιπόν ε, τις εμπορικές συναλλαγές με την γύρανση, γιατί υπάρχει επίδραση από την γύρανση του πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο και πρέπει και τέτοιου είδους ζητήματα να απαντηθούν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες δείκτες και για αυτά. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπεσέ. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Συνάδελφοι, μόλις ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Όχι, κύριε Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για να κλείσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Κάπως έντονη θα έλεγα, αλλά πάντως στα όρια της αυρότητας. Θα ήθελα να πω ότι εδώ το, ζητούμενο, το ζήτημα μάλλον δεν είναι τώρα να κάνεις πράσινο σημείο. Το θέμα είναι να ξέρουμε, να έχουμε μια ορθολογιστική προσέγγιση και να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η, πραγματικότητα που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια ακόμα. Ο κόσμος, ο κόσμος αλλάζει κύριε Πίπερ. Και αφού αλλάζει ο κόσμος πρέπει να αλλάξουμε και γυαλιά. Άλλωστε, το ζήτημα αυτό των δικτών, συμπληρωματικών ως προ το ΑΕΠ δικτών, είναι κάτι όχι το ευρωπαϊκό μόνο, δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά είναι κάτι που συζητούν σε ολόκληρο τον κόσμο όλα τα σοβαρά οικονομικά ερευνητικά κέντρα ε, και πρέπει να σας πω ότι εγώ από τη Γαλλία, την πατρίδα μου, έχω τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι ακριβώς ο καλύτερος φίλος των Πρασίνων ο οποίος θέσπισε μια ε, μονάδα κοινωνικών μελετών με επικεφαλή τον κύριο Στίγκλιτς, ε, Αμερικανό οικονομολόγο, για να εξετάσει αυτούς τους δείκτες. Και ναι, το συζήτησαν, το μελέτησαν πολλοί άνθρωποι αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορεί τα πράγματα να είναι η εικόνα που Μα δίνουν κάποιοι δείκτε μπορεί να είναι και αντιφατικοί ακόμη πολύ περίπλοκοι σε ορισμένου τομεί. Άλλωστε αυτό ισχύει και για το ΑΕΠ, ειδικά στην αρχή. Το ΑΕΠ μα έδινε πολύ στρεβλωμένη εικόνα για ορισμένα πράγματα ε, και όμω μετά σιγά σιγά διορθώθηκε και όπω είπε και η Επιτροπή έχει αλλάξει η κατάσταση στου δείκτε αυτού. Υπάρχουν κάποιε απλέ ενδείξει. το μόνο που χρειάζεται είναι να τους συνενώνουμε, να κάνουμε δηλαδή την κατάλληλη τον κατάλληλο συνδυασμό των δικτών αυτών και όπως υπόθηκε και νωρίτερα υπογραμμίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα ε, απάλληψης του ΑΕΠ ως κύριου δίκτυ. Υπάρχει γιατί είναι ο δίκτυς ο οποίος προσμετρά την οικονομική ανάπτυξη, αποτελεί τον τρόπο υπολογισμού του, οικονομικού πυλώνα της ανάπτυξής μας, της κοινωνίας μας. Ε, αυτό που λέμε σωστικά είναι ότι ο οικονομικός πυλώνας δεν αρκεί για να δούμε αν είμαστε καλά, αν πάμε καλά. Υπάρχει και ο κοινωνικός, υπάρχει και ο περιβαλλοντικός πυλώνας, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον οικονομικό. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέσα για να ε, εξετάσουμε το δυναμισμό αυτό, τη συμπληρωματικότητα και την ε, συνεργατική ε, σχέση, την εταιρική σχέση μεταξύ των τριών αυτών πυλώνων. Και γι' αυτό ακριβώς και στην γνωμοδότηση που σας έχω υποβάλει προς έγκριση λέμε ότι ε, το ΑΕΠ ε, ως μέτρο υπολογισμού μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια απαραίτητη αναφορά για την εκτίμηση ανάπτυξης των περιφερειών κτλ. Αλλά ανεπαρκή απαραίτητη αλλά ανεπαρκή. Και βεβαίως θα πρέπει να ε, ακούσουμε τους ειδικού γι' αυτό και θα συμφωνήσω κι εγώ με την πρόταση για μια ακρόαση, μια συνάντηση εδώ. Καλή πρόταση να μπορέσουμε να ενημερωθούμε κι εμείς ε, και να φτάσουν, να έχουμε την πιο επίκαιρη ενημέρωση πάνω απ' όλα. Αλλά θέλουμε με την γνωμοδότηση αυτή να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τι εργασίε για την επικαιροποίηση αυτών των δικτών. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυροπεμένα και να περιμένουμε να μα πέσει ο ουρανό στο κεφάλι. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίε, πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε αυτά τα πολιτικά μηνύματα, τα σαφή πολιτικά μηνύματα κατά τρόπο ουσιαστικό και θετικό. Ευχαριστώ. Νομίζω ο κύριος το, το Έλερ κάτι θέλησε να πει ε, χωρίς να ξαναλύγει συζήτηση, απλώ ε, σας ξέχασα νωρίτερα, ο κύριο Τσέλερ. Ναι, Πρόεδρε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να λάβω εγώ το λόγο αφού έχει κλείσει ο εισηγητή, ο συντάκτη τη νομοδότηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω ότι βεβαίω μπορούμε να συζητούμε εάν μπορούμε με του δείκτε πέραν του ΑΕΠ να περιγράψουμε καλύτερα τη συνθήκη ζωή ε, από ότι το ΑΕΠ. Ασφαλώ θα υπάρχουν τέτοιου είδου δείκτε και ασφαλώ, υπάρχει και μια πληθώρα προτάσεων για το πώ μπορούμε αυτού του δείκτε να του ε, χαρακτηρίσουμε, είτε πρόκειται για κοινωνική, είτε πρόκειται για περιβάλλον, είτε πρόκειται για ποιότητα ζωή, είτε πρόκειται για έρευνα, για κοινωνική ε, ισότητα, ε, εκπαίδευση, ευκαιρι... ισότητα ευκαιριών κτλ. Μια σειρά δικτών υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώ θα του αξιοποιήσουμε, πώ θα του κρίνουμε. Το έθιξε και η κυρία Κρέλ νωρίτερα. Είναι συγκρίσιμοι αυτοί οι δείκτε από το ένα κράτο στο άλλο και άλλωστε πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολύ διαφορετικέ συνθήκε, όχι μόνο από κράτο σε κράτο, αλλά μεταξύ διαφόρων περιφερειών του ίδιου κράτου μέλου. Πώ θα του περιγράψουμε λοιπόν του δείκτε αυτού. Και επίση ο τρόπο με τον οποίο διεξήχθη τώρα ακριβώ συζήτηση είναι ε, αφήνει αυτό το ζήτημα το πώ χειριζόμαστε από εδώ και μπρος την κοινωνική πολιτική, την ε, πολιτική συνοχή, την περιφερειακή πολιτική. Ε, υπάρχει ζήτημα δηλαδή να εγκαταληφθεί η πολιτική συνοχή και να προχωρήσουμε προς νέες τάσεις, προς νέους προσδορισμούς. Εδώ δηλαδή αφήνουμε τα ταμεία που έχουμε μέχρι τώρα και που εξυπηρετούν εδώ και χρόνια του στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής, περιφερειακή πολιτική μεταφορών και ό,τι άλλο, ε, διότι θεωρούμε ότι μπορούμε με διαφορετική κατάταξη, κατανομή, να εξασφαλίσουμε καλύτερα τους στόχους μας. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι ε, εγκαταλείπουμε την περιφερειακή πολιτική σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική συνοχή, η στρατιωτική πολιτική έχει απόλυτη σημασία ακόμη και τώρα για την ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουμε να κάνουμε βεβαίω με κάποια προβλήματα που πρέπει να διαγνώσουμε, δηλαδή καθυστέρηση ανάπτυξη σε, κάποιους, σε κάποιε περιφέρειε τη Ευρώπη που πρέπει να διαγνώσουμε με τον σωστό τρόπο. Αλλά εδώ θα ήθελα εγώ να προσθέσω ότι οι περιφέρειε ίδιε είναι αυτέ που ξέρουν καλύτερα τι χρειάζονται και πού χρειάζονται επενδύσει και πώ μπορούν να επενδύσουν καλύτερα τα χρήματα τα οποία μπορεί ενδεχομένω να λάβουν ως στήριξη. Και γι' αυτό χρειάζεται το ΑΕΠ πάντα. Και επίσης ως βάση για την ε, κατανομή των κονδυλίων και για την αναγνώριση της ποιότητας ε, της δραματικής πολιτικής, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ορίσουμε μόνο ένα πλαίσιο και στη συνέχεια, όπως υπόθηκε πολύ ωραία ήδη εδώ, να αφήσουμε σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό δηλαδή επίπεδο, τον προσδιορισμό της χρήσης, του τρόπου χρήσης αυτής της στήριξης που θα προσφέρει το πλαίσιό μας. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτά τα πράγματα να τα ορίσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά τρόπο ομοιόμορφο, επιτόπου, σε τοπικό επίπεδο, ε, εκεί που ενδεχομένως βλέπουμε κάποια δυσκολία. Μία πόλη, ένα χωριό, μια περιφέρεια μπορεί να αποφασίσει μόνο της τι χρειάζεται και πώς. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε άνοφεν. Και επίσης η... Συνθήκες ζωής ε, είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια και ίσως ε, θα χρειαστεί πολύ συζήτηση για να δούμε τι είδους δείκτες χρειαζόμαστε για να τις ε, περιγράψουμε. Και κατά τα άλλα θεωρώ ότι για την πολιτική συνοχή, για την ερωτική πολιτική χρειαζόμαστε τους αποδεδειγμένα καλούς δείκτες, δεν πρέπει δηλαδή να βγούμε από την πεπατημένη. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Σα υπενθυμίζω ότι 29 Νοεμβρίου ε, ψηφίζει η κατ' ουσίαν αρμόδια επιτροπή και ω εκ τούτη γνωμοδότηση δική μα για να ληφθεί υπόψη πρέπει το αργότερο να ψηφιστεί 27-28 Οκτωβρίου από την Επιτροπή περιφερειακής πολιτικής. Θα πρότεινα λοιπόν προθεσμία για τις τροπολογίες την 5η Οκτωβρίου, τις 5 Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι ε, δεδομένου ότι ήταν πολύ ε, διεξοδική η συζήτηση σήμερα, θα είναι πιο εύκολο να ε, συντάξετε και να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Παρακαλώ όμως μη τους χρονικούς περιορισμούς που έχουμε. 5 Οκτωβρίου λοιπόν προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Επίσης έχουμε και δράση μακροπρόθεσμη να προσδιορίσουμε ημερομηνίες για τις ακροάσεις που θέλουμε στις αρχές του 2011. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επί τη ευκαιρία των ακροάσεων αυτών λοιπόν. Και τώρα θα πρότεινα να προχωρήσουμε στην εξέταση της πρότασης για, την, για τις κρατικές ενισχύσεις σε περίπτωση ε, κλεισίματος ε, ανενεργών ανθρακουριχίων και πιστεύω ότι ο κ. Σετίνη θα θέλει να λάβει το λόγο. Για αν έχει το λόγο παρακαλώ. Κύριος Πρεζίνα. Πρόεδρε ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη, εκλήθεν σχετικά βραχυπρόθεσμα και βάλαμε το θέμα αυτό στην τελευταία, στην τελευταία στιγμή στην ημερήσια διάταξη γιατί πρόκειται να γίνει η εξέταση της εκθέσεως στην κατουσία αρμόδια πολιτική ε, επιτροπή ε, πολύ σύντομα και ως εκ τούτου η γνωμοδότησή μου πρέπει να εξεταστεί. Δεν έχουμε να κάνουμε με ε, επιπτώσεις που προκύπτουν από την εκπνοή όλου του νομοθετικού πλέγματος που έχει να κάνει με τη στήριξη ανθρακοριχείων που κλείνουν και που αφορά τη ζωή και την επιβίωση 100.000 πολιτών μας τουλάχιστον. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ανθρακοριχεία Ε, Γερμανία, Ισπανία, Σλοβακία, ε, κατ' ουσίαν είναι οι χώρες που επηρεάζονται από το κλείσιμο των ανθρακοδρυχείων, ε, τα οποία εφόσον δεν είναι για το μέλλον ανταγωνιστικά θα πρέπει να τύχουν κρατικών ενισχύσεων με σημαντικές φυσικά περιφερειακές και οικονομικές επιπτώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η δική μας Επιτροπή να ε, έχει έτοιμη την γνωμοδότησή της. Έχω λοιπόν καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες για την ε, αντιμετώπιση της κατάστασης. Τροπολογία υπαριθμών 4 αναφέρεται στο γεγονός ότι ε, δεν επετεύχθη σε ορισμένες περιπτώσεις η απαραίτητη συνένεση και έτσι Ήδη το 2018 προβλέπεται το κλείσιμο ορισμένων προβλεπόταν μάλλον το κλείσιμο κάποιων ανθρακοριχείων στη Γερμανία και τώρα η Επιτροπή προτείνει το 2014 ε, που όμως ε, είναι πολύ νωρίς πιστεύω θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να ε, βρεθούν, ε, να δοθούν περιθώρια ε, χρονικά στις περιοχές αυτές. Είναι ήδη πολύ νωρίς και πολύ σημαντικές οι οικονομικές επιπτώσεις ε, για τις περιοχές αυτές. Επίσης, τροπολογία υπαριθμών 16 ε, επισημαίνει το κύριο σφάλμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δηλαδή αυτά τα ανθρακοριχεία που θα κλείσουν Ε, αναφέρεται θα έχουν θετική, θετικό αντίκτυπο ως προς τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ όμως γνωρίζω ότι πολλοί είναι οι επιστήμονες που πιστεύουν όπως και εγώ ότι Η καύσιμη ύλη την οποία προσέφεραν αυτά τα ανθρακοριχεία που τώρα κλείνουν θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποια άλλη καύσιμη ύλη καύσιμη και ως εκ τούτου θα έχουμε επιβάρυνση ακόμη ε, μεγαλύτερη από εκπομπές προερχόμενες από τις μεταφορές που θα από τις διαδικασίες μεταφορών που θα χρειαστούν για τη μεταφορά αυτών των νέων καυσίμων ε, υποκατάστασης. Επίσης, τροπολογία 15 αναφέρεται στα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων, ότι δηλαδή χρειάζεται η περιφερειακή πολιτική ε, να εξασφαλίσει λύσεις ε, που θα αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις ε, του κλεισίματος αυτών των ορυχείων. Στη δε τροπολογία 18 προτείνουμε συγκεκριμένες προθεσμίες για το κλείσιμο των θερκορυχείων, δηλαδή τη χρονολογία του 2020. Στην τροπολογία 19 μιλούμε για το ενδεχόμενο να έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι μπορεί ένα ανθρακοριχείο ε, να αντιμετωπίζει σήμερα οικονομικές δυσκολίες, να μην είναι ανταγωνιστικό, αλλά λόγω φερρυπίν πιθανών ε, ανακατανομών ως προς την οικονομική ισχύ των διαφόρων καυσίμων και, τις και δεχόμενων διακυμάνσεων τιμών μεταξύ ε, ε, φυσικού αερίου, πετρελαίου και το καθεξής μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα και ο άνθρακας να καταστεί και πάλι ανταγωνιστικό στα ανθρακοριχεία αυτά εν προκειμένου. Γι' αυτό με την ε, τροπολογία υπαριθμών 19 εισάγουμε μια παρέκκληση στον κανόνα του κλεισίματος το 2020. Να αφήσουμε δηλαδή να ανοιχτή τη δυνατότητα εάν σε ορισμένες και ε, με περιπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά αυτά τα ορυχεία για μια περιοχή, Θέλουμε να, ε, για να ανατραπούν οι συνθήκες θέλουμε να ε, υπάρχει δυνατότητα να μην κλείσουν το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλουν συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Πίπε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Έχουμε εδώ να κάνουμε με το δεδομένο ότι σε ορισμένα κράτη ο άνθρακας δεν είναι όντως ανταγωνιστικός, Ισπανία, Γερμανία κτλ. Αλλά από την άλλη έχουν κάνει επιλογές ε, οι κυβερνήσεις οι οποίες ε, ορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα επαρκές για την αντιμετώπιση των, ε, της, αυτού του προβλήματος ανταγωνιστικότητας, τις οποίες όμως τώρα προθεσμίες περιορίζει ακόμη περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν λοιπόν ξαφνικά υποθεί ότι αντί για... 10 χρόνια προς, ή για 8 χρόνια δίνουμε περιθώριο μόνο 4 χρόνια για να κλείσουν αυτά τα ορυχεία, Προφανώ θα χάσει ο κόσμο την εμπιστοσύνη του στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ο κόσμο από τη Μαδρίτη ή από το Βερολίνο θα αντιδράσουν στην ίδια την Ευρώπη γιατί θα δουν ότι είναι ακόμη πιο δυσμενή η συμπεριφορά τη σε σχέση με τι εθνικέ κυβερνήσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις που ουσιαστικά έχουν ληφθεί. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο για ε, ορυχεία τα οποία παραμένουν ανταγωνιστικά. Εκεί θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάποιες από τις συνθήκες, αλλά για τα μη ανταγωνιστικά αυτά που πρέπει να κλείσουν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Και ευχαριστώ επί τη ευκαιρία για την υποστήριξη και τον κύριο Μπρεζίνα όλος ιδιαίτερος. Ο κύριος Λάστρα δεν ξέρω αν θέλει κανείς μετά να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο βασικά αφορά τέσσερις χώρες, αλλά είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αφορά πάνω από 100.000 ε, θέσεις απασχόλησης, μπορεί να υπάρχει λοιπόν κοινωνικός αντίκτυπος ιδιαίτερα σοβαρός ε, και το κλείσιμο των ανθρακοριχείων αυτών ε, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Νομίζω ότι η ημερομηνία 2014 είναι εντελώς αυθαίρετη τυχαία και χρειαζόμαστε μια ημερομηνία εκπνοής ε, που να πηγαίνει μέχρι το 2018, ενδεχομένως μέχρι και το 2020. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, οι συνέπειες στις ε, διάφορες χώρες. Δύο βασικά στοιχεία θα ήθελα να τονίσω, ειδικότερα όσον αφορά τον άνθρακα και την εξόριξη. Έχουμε μία περιβαλλοντική πτυχή. Ο άνθρακας ε, θα ε, αντικατασταθεί από άλλης προέλευσης ε, άνθρακα και ενδεχομένως τα επίπεδα μόλυνσης να διατηρηθούν. Δεν ξέρω, ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούσε να μας πει τι προτίθεται να κάνει γι' αυτό. Όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα, έχουμε και ένα νέο σενάριο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι υπάρχουν 12 προγράμματα πιλωτικά που αφορούν την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τα ανθρακοριχεία πιο αηφόρα, πιο ανταγωνιστικά και επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε προκειμένου να ε, μην ρηπαίνουν τόσο πολύ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν ενισχύσεις του τύπου, για παράδειγμα, της βιομηχανίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ε, πάνω από 100.000 άτομα ε, αφορά το ζήτημα αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους και νομίζω ότι ό,τι και να γίνει θα έπρεπε να παρατείνουμε λίγο την ημερομηνία του 2014. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να την αναβάλουμε μέχρι το 2018-2020. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vieles ist ja von den Kollegen bereits. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το έθιξε μόλις ο συνάδελφος. Πολλά είναι τα σοβαρά επιχειρήματα για τα οποία οι λύσεις που έχουν ε, ήδη προσδιοριστεί σε επίπεδο Ευρωπα... Ε, κρατών μελών για ένα ε, πλαισιωμένο τρόπο κλεισίματος, μια διαδικασία πλαισιωμένη κλεισίματος αυτών των ε, ε, ανθρακοριχείων δεν θα πρέπει να ανατραπούν από την Ευρωπαϊκή πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως και να μην ε, βάζουμε τρικροποδιές στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη και ανάπτυξη των, στις, και των νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και της σύλληψη και συγκράτησης άνθρακα και βεβαίως θέλουμε πάνω από όλα, αν έχω αντιληφθεί σωστά την κατάσταση, να ορίσουμε χρονοδιαγράμματα ανεκτά βιώσιμα. Δεν μας ενδιαφέρει να χρηματοδοτήσουμε παόριστον τα μη ανταγωνιστικά ανθρακοριχεία. Όχι. Και δεύτερον, δεν θέτουμε να αμφιβόλο τις προσπάθειες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων. Γι' αυτό παρακαλώ την ε, τροπολογία 9 να την αντιληφθείτε ως τέτοια. Δεν θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει κάποια παρεξήγηση λόγω του κειμένου που υπάρχει. Μάλιστα, κ. Μπριζίνα θα ήθελα και πάλι να συνοψίσει. Για την τροπολογία 9 θα ήθελα να επιμείνω. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τον κλιματικό αντίκτυπο της παραγωγής άνθρακα, της καύσης του άνθρακα, ε, στις ε, εγκαταστάσεις ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχω δει πολλές φορές τέτοιες εγκαταστάσεις. Έχω περάσει πολλά χρόνια εγώ ίδιος ως ανθρακορίχος και γνωρίζω, ξέρω γιατί μιλάω. Όμως ε, ο άνθρακας αυτός θα αντικατασταθεί από άνθρακα που θα εξορίσεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς ε, είναι μηδενικός ο αντίκτυπος ε, σε οποιαδήποτε αλλαγή του κλίματος ως προς την εκπομπή των αερίων. Γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να μεταφερθεί αυτός ο άνθρακας, για παράδειγμα, από την Αυστραλία, που είναι πολύ φθηνός παρεμπιπτόντος. Οπότε στην περίπτωση της Ισπανίας ε, νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο ισπανικός άνθρακας θα αντικατασταθεί από τα, τον άνθρακα της Αυστραλίας ε, που θα εισάγεται μέσω των ισπανικών λιμένων. Οπότε δεν είναι θέμα αμφιβολιών ε, για τον μηδενικό αντίκτυπο. Αν υπάρχει όμως οποιαδήποτε αντίρρηση, ευχαρίστω να, την να την αποδεχθώ. Πρόεδρο, ναι, βεβαίω θα υπάρξει και χρόνος για περαιτέρω διευκρινήσει, γιατί έχουμε ούτω ή άλλω ε, προθεσμία μέχρι τι 8 ε, Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι για τις τροπολογίες. Παρακαλώ να σεβαστείτε την προθεσμία αυτή. Μέχρι τότε ελπίζω να έχουμε και τι μεταφράσει. Θα ήθελα να προτείνω όμω να μην περιμένουμε. μεταξύ δηλαδή να επεξεργαστούμε τις ε, τροπολογίες. Ο μόνος τρόπος να φτάσουμε στην Οικονομική Επιτροπή πριν από την ψηφοφορία εκείνη ε, της 9ης Νοεμβρίου είναι να ψηφίσουμε εδώ 27-28 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 14. Η κυρία ε, Λένα Κολάσκα Μπομπίνσκα είναι η συντάκτρια τη γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του σχεδίου δράση για την ενεργειακή απόδοση. Και θα ήθελα να ζητήσω από τη Λένα να παρουσιάσει το ζήτημα. Dziękuję bardzo. Właściwie to e, ja wolałabym, żeby pani jako przewodnicząca. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την έκθεση αυτή, κυρία Πρόεδρε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι εγώ πρέπει να συντάξω μια γνωμοδότηση. Αλλά ήθελα εσείς πρώτα απ' όλα να μας πείτε ποιες είναι οι προθεσμίες. Ε, υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και από άποψη διοργάνωση, ώστε εγώ δεν ξέρω πλέον τι να κάνω. Πρέπει να τη γράψω τη γνωμοδότηση, δεν πρέπει να τη συντάξω. Τι ακριβώς θα γίνει. σε κάθε περίπτωση εγώ έχω δουλέψει, ο κύριος Πίπερ έχει στείλει τις τροπολογίες του αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν θα υποβληθεί τελικά η γνωμοδότηση αυτή ή όχι. Για πείτε μου. Πρόεδρος. Πράγματι υπάρχει μια αβεβαιότητα που δεν οφείλεται σε εμά τους ίδιους. Είναι αβεβαιότητα που οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή Ήτρε δεν μας έχει επισήμως ανακοινώσει εάν θα αναβάλει την ψηφοφορία του δικού τους εγγράφου, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ όσων κατάλαβα, έχει αναλάβει τη δική της ψηφοφορία, την έγκριση δηλαδή των δικών της αντιστοίχως κειμένων. Πάντως, μάλλον θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει την γνωμοδότηση αυτή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, γιατί η Ήτρε μάλλον θα διατηρήσει τις προθεσμίες του Νοεμβρίου. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε βάσει αυτής της εικασίας, πρέπει να εργαστούμε βάσει της υπόθεσης ότι θα ε, ε, χρειαστεί αυτή η γνωμοδότηση. Εάν δεν χρειαστεί, Θα σας καλέσω να αποστείλετε απευθείας τις τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή της εδώ γνωμοδότησης στην Επιτροπή Ήτρε. Και στις 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση σχετικά στο Στρασβούργο. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί σε όλες τις δυνατότητες προς στιγμή. Πάντως πρώτη μας επιλογή προφανώς είναι η γνωμοδότηση αυτή και να προωθηθεί και να την εγκρίνουμε. Ιδάλλως θα πρέπει να την μετατρέψουμε σε τροπολογίες που θα υποβάλουμε αμέσως ως ε, τροπολογίες της έκθεσης της Επιτροπής Ήτρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω ετοιμάσει πέντε σημεία στα οποία ήθελα να σταθώ για την παρέμβασή μου. Πρώτα απ' όλα, βεβαίως, η περιφερειακή συνιστόσα είναι πιο σημαντική. Υπάρχουν πολλές εντάσεις, αψημαχίες και συζητήσεις σχέση με την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους λοιπόν ή όχι. Αυτό είναι ήδη ένα σημείο που έχει προκαλέσει θερμή συζήτηση. Στο ΕΛΚ συζητήθηκε, σε όλες τις διαπραγματεύσεις επανέρχεται, είναι σημαντικό για όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν πολύ ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η συμβαστική πρόταση που θα εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση Έχουμε μελετήσει τις λεπτομέρειες του ζητήματο αυτού, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στα περιφερειακά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αποκέντρωση για σκοπούς ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα πρέπει να υπάρξει πολυεπίπεδη διοργάνωση και να ξαναδούμε από άλλη άποψη την ενεργειακή αποδοτικότητα, να σκεφτούμε την έννοια του smart cities, των ευφυών πόλεων. Έπειτα, λέμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη το πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά σε επίπεδο περιφερειών. Διότι υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις από τη μια στην άλλη περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Δεν θα πρέπει μια κεντρική προσέγγιση να επιβάλλεται άνωθεν. Αυτά ε, είναι έτσι αλλιώ πράγματα που τα αναλύει το κείμενό μου, δεν θα μπω εγώ στι λεπτομέρειε. Ο κύριο Πίπερ έχει υποβάλει μια τροπολογία. Θα την ε, υποβάλω, θα την, εγκρι... θα την υιοθετήσω και ω δική μου, οπότε θα την υποβάλω και εξ ονόματό μου. Και λέγεται ότι θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που να προσεγγίζει τις απαιτήσεις της οδηγίας για την οικολογικό σχεδιασμό και την ετικετοθεσία. Έχουμε πολλές διατάξεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα σε αυτό το κείμενο. Δεν χρειάζεται τώρα να χαθούμε προσπαθώντας να εξεύρουμε νέες λύσεις εκ του μηδενός. Θα πρέπει να βασιστούμε στις λύσεις που ήδη υπάρχουν και προβλέπονται. Εδώ μιλώ για όλον τον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αλλά βεβαίως αυτό πρωτίστως είναι σημαντικό για τη δική μας την Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε νέε διατάξει ούτε νέου κανόνε με το κείμενό μα, αλλά να βασιστούμε σε λύσει που ήδη υπάρχουν. Και θα πρέπει λιγάκι να επιταχύνουμε του ρυθμού μα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλε αυτέ τι ιδέε μα όταν το δυνατόν συντομότερα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ήθελε κάποιο να συμπληρώσει όσα μόλι υπόθεταν. Από την κυρία Κολάρσκα Μπουμπίνσκα. Όχι, δεν υπάρχουν σχόλια. Να σα ζητήσω λοιπόν να σεβαστείτε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, όπω και στι προηγούμενε περιπτώσει, είναι 8η Οκτωβρίου το μεσημέρι. Επίση, ελπίζουμε οι μεταφράσει να φτάσουν στα χέρια μα πριν την λήξη τη προθεσμία τη τροπολογία. Σα ενθαρρύνω θερμά να διαβάσετε προσεκτικά την έκθεση και να την μελετήσετε. Η περιφερειακή πολιτική έχει συμβάλει ιδιαιτέρως στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι λοιπόν αυτό σημαντικό και για το μέλλον, γιατί θα πρέπει η πολιτική μας να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο να επηρεάζει. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν σχόλια, 8 Οκτωβρίου το μεσημέρι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στο 15, στα διάφορα, δεν έχω εγώ τίποτε άλλο να προσθέσω. στο 16 να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 4 Οκτωβρίου Δευτέρα, η ημέρα των ανοιχτών πορτών. Σας ενθαρρύνω όλους να παρευρεθείτε σε δύο εκδηλώσεις τουλάχιστον στις ανοιχτές πόρτες. Πρώτα απ' όλα η εναρκτήρια συνεδρίαση, θα έχουμε περίπου μία ώρα για συζήτηση στο ημικύκλιο και έπειτα ακόμα μια συνάντηση όπου θα είμαστε εμείς και η Επιτροπή Κοτέρ της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα συνσυνεδριάσουμε λοιπόν στις 5 Οκτωβρίου, Τρίτη στις 9 το πρωί συγκεκριμένα. Συζήτηση για την πολιτική συνοχής και τη στρατηγική 2020. Ελπίζω λοιπόν να σας δω εκεί. Και έπειτα έχουμε Εκατοντάδε εκδηλώσει την ημέρα των ανοιχτών, την εβδομάδα των ανοιχτών πορτών, υπάρχουν σεμινάρια, ομιλίε, πάρα πολλά που θα γίνουν. Ελπίζω λοιπόν να φροντίσετε να είμαστε κι εμεί αρκετά ορατοί και να προβάλλουμε τι εργασίε μα σε αυτέ τι συναντήσεις. Τελευταία επισήμανση ήταν αυτή για την μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να θέσετε, έληξε η συνεδρίασή μα. Ευχαριστώ.